Ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τώρα τον δόκτορα Αλή Αμπντέλ Αλ Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αραβικής Δημοκρατίας ε, της Αιγύπτου, ε, που συνοδεύεται και από ε, μια πολύ σημαντική αντιπροσωπεία από τον πρέσβη κ. Χαλή Αμπτελάλα. Ε, κύριε Αλή Αμπτέλ Άλε, είναι πολύ έγκαιρη η προσέλευσή σας ε, στην ε, συνεδρίασή μας. Πρέπει να σας πω ότι εμείς θέλουμε και αξιολογούμε πολύ θετικά την σταθερότητα της χώρας. Ο κύριος Μουστάφα Αλ Μαγκούλη είναι η πρώτη περίπτωση σημαντικής αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει και ε, γυναίκες. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση για την ε, ασφάλεια, γνωρίζουμε ότι 70% των Αιγυπτιακών στρατευμάτων αποσύρονται από την Χερσόνησο του Σινά. Θα θέλαμε όμως να μας δώσετε τις δικές σας απόψεις ε, και να μας δώσετε και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή καθώς επίσης και τις σχέσεις με τη Λιβύη και με την Γάζα. Επίσης, ε, στην Ένωση της ε, Μεσογείου κατέχετε την θέση του Προέδρου ε, και γνωρίζουμε ότι έχετε συζητήσει χθε με τον Πρόεδρο Ταγιάννη για θέματα τα οποία αφορούν την Μεσόγειο. Θα να μας πληροφορήσετε και γι' αυτό. Στα πλαίσια της συνεργασίας ε, μεταξύ των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Αιγύπτου που ενδυναμώθηκαν από την απόφαση συνεργασίας του Ιουλίου του 2017 τα πράγματα ευελπιστούμε ότι θα και οι σχέσεις θα ενταθούν ακόμα περισσότερο. Επίσης θα θέλαμε να μας πείτε και δύο λόγια σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας στην Αίγυπτο θέλουμε να μας διαβεβαιώσετε για, την, για τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι ε, αυτή η αναφορά θα είναι σαφής στο Αιγυπτιακό Σύνταγμα. Ε, αγαπητέ Δόκτωρ Αλή Αμπτελ Άλλα, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Μακάλιστερ, ε, Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. You can speak in whichever language you wish. Μπορείτε να μιλήσετε όποια γλώσσα θέλετε, λέει ο πρόεδρος. Θα υπάρχει όμως διερμηνία. Somebody to, to do the translation in English. Okay, then we'll go ahead. We'll go ahead. Okay. Voilà, c'est toujours le problème voilà, de la traduction. Υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα μετάφρασης αλλά το σημαντικό είναι να μιλήσει κανείς μία γλώσσα η οποία θα γίνει κατανοητή από όλους. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα προσπαθήσω ε, να μιλήσω στα ε, γαλλικά. Και ευελπιστώ ότι και από τα γαλλικά θα υπάρξει μετάφραση προς όλες τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μακάλιστερ τον πρόεδρο του, ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος ε, του, της Βουλής ε, της Αιγύπτου ε, επισκέπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το 2004. Η κατάσταση στην Αίγυπτο και από την 30 Ιουνίου του 2013 έχει αλλάξει. Υπάρχει ένα νέο σύνταγμα, ένας νέος πρόεδρος και επίσης μια νέα βουλή. Το κοινοβούλιο μας στην Αίγυπτο αποτελείται από 596 βουλευτές. Όχι, ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ρωτά ο, ο πρόεδρος της Βουλής, ε, γιατί βλέπω ότι σηκώνουν διάφορα τα χέρια τους. Ε, απλώς θέλουν, λέει ο πρόεδρος, να πάρουν το λόγο. Νόμιζα ότι κάτι λέω που δεν τους ικανοποιεί. Γι' αυτό σταμάτησα, λέει ο πρόεδρος της Βουλής της Αιγύπτου. Έχουμε λοιπόν 90 γυναίκες βουλευτές, 39 ε, κόπτες ε, και 20 πολιτικά κόμματα. Η πλειοψηφία στο Βουλή της Αιγύπτου ε, αποτελείται από συνασπισμό ε, πολλών βουλευτών που προέρχονται από κόμματα αλλά και ανεξαρτήτων βουλευτών. Έχουμε δουλέψει σε, πάνω σε πολλά νομοσχέδια ε, ε, στην χώρα μου, έτσι ώστε να εξυγχρονίσουμε ε, την Αίγυπτο από κοινωνικής και οικονομικής πλευράς. Έχουμε περάσει περίπου 400 νόμους μέσα σε τρία χρόνια. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και νόμοι ιδιαίτερως σημαντικοί που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της αρχής της ισότητας ε, ε, όλων των Αιγυπτίων και κυρίως ε, της ισότητας ανάμεσα στους μουσουλμάνους και τους κόπτες. Έχουμε Έχουμε νόμους που αφορούν ακριβώς την δημιουργία εκκλησιών και την κατασκευή εκκλησιών. Βάσει των νόμων αυτών και οι εκκλησίες και τα τεμένη, τα τζαμιά, ε, ε, οικοδομούνται βάσει ενός και μόνο κανόνα. Δηλαδή, μια εκκλησία που θα υπόκειται στους ίδιους νόμους, είτε πρόκειται για κοπτική εκκλησία είτε πρόκειται για τέμενος. Πρόκειται για ε, ε, νόμους ε, οι οποίοι ενισχύουν λοιπόν την έννοια της ισότητας των Αιγυπτίων πολιτών. Είχαμε και έναν άλλο νόμο που αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Η πλειοψηφία των πολιτών στην Αίγυπτο δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες ε, για να πάει στο νοσοκομείο ε, ή για να χρησιμοποιήσει άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Βάσει όμως αυτού του νόμου, κάθε Αιγύπτιος, όπως και κάθε Ευρωπαίος, πληρώνει, κάθε Αιγύπτιος λοιπόν λέω, πληρώνει μία εισφορά, έτσι ώστε να έχει δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε και έναν άλλο νόμο που αφορά τις επενδύσεις στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με αυτόν τον επενδυτικό νόμο, λοιπόν, οι επενδύσεις πλέον απελευθερώνονται. Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής μπορεί να μεταφέρει χρήματα στην Αίγυπτο για να οργυρώσει το σχέδιό του και έχει δικαίωμα να μεταφέρει τα κέρδη από την Αίγυπτο προς το εξωτερικό ελεύθερα. Στο νόμο αυτό λαμβάνονται υπόψη και οι διεθνείς ε, συμφωνίες προστασίας και οι διεθνείς ρυθμίσεις προστασίας των ξένων επενδύσεων. δεν υπάρχουν ενθυκλοποιήσεις, δεν υπάρχουν κατασχέσεις και επομένως αντιθέτως ε, ε, παρέχονται εγγυήσει για τους ξένους επενδυτές που θα αποφασίσουν πλέον να επενδύσουν στην Αίγυπτο. Υπάρχει άλλος ένας νόμος που αφορά την ελευθεροτυπία. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, σαφώς ε, απαγορεύεται να φυλακιστεί δημοσιογράφος ε, ε, λόγω των όσων έχει γράψει στον έντυπο τύπο ή σε όσα έχει πει στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. Διασφαλίζεται λοιπόν η ελευθερία έκφρασης. αυτή οι νόμοι που ανέφερα ε, είναι θεμελιώδους σημασία στην Αίγυπτο. Υπάρχουν όμως και άλλοι νόμοι που ε, αφορούν όλες τις οικονομικές και κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της ε, ζωής. Η κατάσταση στην Αίγυπτο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι συγκεκριμένη. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Η πρώτη πρόκληση αφορά βέβαια την τρομοκρατία. Δεύτερη πρόκληση είναι το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης. Και υπάρχει και ένα τρίτο πρόβλημα που μια μεγάλη πρόκληση ε, που είναι η οικονομική κατάσταση. Όσον αφορά την τρομοκρατία ε, που συνδέεται άμεσα και με το δεύτερο πρόβλημα της παράτυπης ε, μετανάστευσης. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά για την τρομοκρατία με τους φίλους ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα είπαμε και χτες με τον Πρόεδρο. Και μάλιστα ο Πρόεδρος της ε, ε, Επιτροπής Άμυνας, αλλά και άλλοι συνάδελφοί σας με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή και έχω μιλήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά και τους λέω πάντα ότι ότι από το 1981 έχουμε πρόβλημα τρομοκρατίας στην Αίγυπτο. Από την εποχή λοιπόν ε, που ο πρόεδρος Αντάτ δολοφονήθηκε από φανατικούς ε, μουσουλμάνους εντός εισαγωγικών των μουσουλμάνους. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν και μετά ξεκίνησε η τρομοκρατία στην Αίγυπτο που σιγά σιγά ε, διονγκώθηκε και πλέον απέκτησε ε, διεθνείς διαστάσεις. Για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία χρειάζεται διεθνής βούληση, δηλαδή όλα τα κράτη θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε από κοινού να βρουν μια λύση για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο, το πρόβλημα του τουρισμού. Συνεργασία ε, κυρίως όσον αφορά την μεταφορά χρηματικών ποσών. Η μεταφορά χρημάτων θα πρέπει να ελέγχεται και αυτό από κάθε χώρα. και κυρίως όσον αφορά ε, και οργανώσεις της κοινωνίας των ε, πολιτών. Είναι σημαντικό να έχουν χρήματα οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά πρέπει να παρακολουθούνται τα χρήματα αυτά. Ε, δηλαδή θα πρέπει ε, κυρίως να διέπονται ε, τα πάντα από διαφάνεια. Θα πρέπει δηλαδή κάθε οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών να δηλώνει από πού προέρχονται τα χρήματα και πού ξοδεύονται τα χρήματα. Γιατί εμείς έχουμε προβλήματα στην Αίγυπτο. Υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες συλλέγουν χρήματα μέσα από εράνους που κάνουν στο δρόμο. Γιατί λένε ότι θέλουν να κατασκευάσουν, ε, να οικοδομήσουν ένα τέμενος ή ένα σχολείο ή ένα νοσοκομείο. Αλλά στην ουσία και στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα είναι ότι, η πραγματικότητα είναι ότι χρησιμοποιούν αυτό το μέσο έτσι ώστε να συλλέξουν χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για τελείως διαφορετικούς σκοπούς. Δηλαδή να χρηματοδοτήσουν τρομοκρατικές ενέργειες είτε στην Αίγυπτο είτε και αλλού. Επομένως, τα κράτη θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να συνεργαστούν έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν τον, ε, την τρομοκρατία. Και θα το κάνουν, θα το καταφέρουν αυτό εάν καταφέρουν να ελέγξουν την κυκλοφορία του χρήματος. Επίπης, επίσης όλα τα κράτη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Μέχρι τώρα, ακόμα και τώρα δηλαδή, υπάρχουν χώρες στις οποίες η Αίγυπτος δίνει πληροφορίες όσον αφορά τρομοκρατικές επιχειρήσεις ή όσον αφορά συγκεκριμένα άτομα που έχουν ε, που θεωρούνται τρομοκράτες ή είναι καταγεγραμμένοι ως τρομοκράτες ε, ε, στις χώρες προέλευσης. και επομένως ε, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και μεταξύ της Αμερικής και μεταξύ της Ευρώπης και μεταξύ των αραβικών χωρών όσον αφορά τι πληροφορίες αυτέ. Επίσης, συνεργασία θα πρέπει να υπάρξει όσον αφορά τον τύπο. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, εφημερίδες και κάποια τηλεοπτικά προγράμματα και κάποια τηλεοπτικά κανάλια τα οποία προωθούν ε, τον, την τρομοκρατία. Υπάρχουν ε, δε κάποια κανάλια τα οποία, ε, τα οποία λειτουργούν στην Ευρώπη και από την Ευρώπη μεταδίδουν τα προγράμματά τους. Τεράστια ευθύνη έχει και η Αίγυπτος όσον αφορά το θέμα αυτό. Και μάλιστα Ναι, πρέπει να σας τα πω όλα αυτά, γιατί η κατάσταση όσον αφορά την δρομοκρατία και την ε, παράτυπη μετανάστευση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Επομένως, πρέπει να σας τα πω όλα αυτά. Η τρομοκρατία λοιπόν έλεγα ότι είναι το, ε, το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα αφορά την παράτυπη μετανάστευση. Η, η Αιγυπτός καταβάλει τρομερές προσπάθειες έτσι ώστε να συγκρατήσει την παράτυπη μετανάστευση. Από τον Σεπτέμβριο του 2007 κα, κανένας μετανάστης και κανένα πλοίο δεν έχει φύγει από την Αιγυπτιακή επικράτεια προς την Ευρώπη. Δεν υπάρχουν ε, δεν υπάρχουν Αιγύπτιοι δε ε, οι οποίοι να βοηθούν αυτή τη διαδικασία ε, αλλά υπάρχουν υπήκοοι άλλων χωρών που προσπαθούν να διευκολύνουν την διάβαση των μεταναστών από την Αίγυπτο. Εμείς στην Αίγυπτο όμως κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να ελέγξουμε το φαινόμενο αυτό. Η σταθερότητα της Αιγύπτου εξαρτάται και από την σταθερότητα της Ευρώπης. Δηλαδή, εάν, ε, μάλλον το αντίθετο, εάν ε, έχουμε ε, και διασφαλίσουμε τη σταθερότητα στην Αίγυπτο, θα υπάρχει σταθερότητα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό ζητούμε από τους Ευρωπαίους φίλους και κυρίως ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσετε έτσι ώστε να ενισχυθεί η χώρα, να ενισχυθεί ε, η ε, κοινωνία της Αιγύπτου, να ενισχυθεί η περιοχή ε, της Μέσης Ανατολής, γιατί οι διαμάχες είναι πολλές, τα προβλήματα και οι σειράξεις είναι πολλές. Έχουμε τη Συρία, έχουμε τη Λιβύη, έχουμε την Ιεμένη, έχουμε το Ιράκ, το Σουδάν, τη Σομαλία κλπ. λόγω ακριβώς αυτών των ε, σειράξεων στην Αίγυπτο έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια ε, μεταναστών που ζουν ε, στο που στην Αίγυπτο. Μεταξύ αυτών 700.000 είναι μόνο οι Σύριοι. Εγώ ε, προσπαθώ να σας δώσω μια γενική έποψη για την κατάσταση στην ε, Αίγυπτο και θέλω να δραχτώ της ευκαιρίας που μου δίνεται η παρουσία μου εδώ έτσι ώστε να συζητήσω μαζί σας ε, αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε και σε κάποια κοινά σημεία και συμπεράσματα γιατί υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Είναι πολλά τα πεδία ε, ε, τα οποία προσφέρονται για συνεργασία ε, και για την κατάσταση στην Αίγυπτο και για την κατάσταση στην, στην Μέση Ανατολή και για την κατάσταση στη Γάζα. γιατί πραγματικά τώρα είναι η στιγμή ε, για να εκμεταλλευτούμε τις πρόοδους που έχουμε κάνει τα δύο τελευταία χρόνια. Και βεβαίως εμείς πάντα βασιζόμαστε ε, στους Ευρωπαίους φίλους ε, έτσι ώστε να παράσχουν βοήθεια. Και για θέματα ε, ελευθερίας του τύπου και για θέματα κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να συζητιούνται όλα τα θέματα αυτά ανοιχτά. Και όλοι μαζί θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτός να σας ακούσω, να συζητήσω μαζί σας ε, και να προσπαθήσω να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις σας ή ε, να ανακουφίσω ενδεχομένως κάποιους προβληματισμού σας όσον αφορά την Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ όλους κύριοι βουλευτές που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν ζητήσει το λόγο οκτώ συνάδελφοι. Η κυρία Λοχμπίλα προστίθεται, άρα εννέα. Επειδή όμως ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όλους, ε, πρέπει βέβαια να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμά μας. Θα έλεγα ε, ο χρόνος παρέμβασης να είναι ένα λεπτό για κάθε ένα από εσάς ε, να καθυστερήσουμε μετά κατά το μέγιστο 10 λεπτά για τη συζήτησή μας με τον επόμενο μιλητή, τον ε, κύριο ε, το Σέχη του Κατάρ. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήλθατε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Είναι κοινέ οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, η μετανάστευση, η τρομοκρατία, ε, σε συνθήκες που είναι όλο και πιο μεταβλητές και όλο και πιο περίπλοκες. Η Αίγυπτος είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πολύ σημαντικός εταίρος και η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι προτεραιότητα για μας. Ανέκαθεν το πιστεύαμε αυτό στη δική μας πολιτική ομάδα. Θέλουμε να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας σε αυτή τη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης και επιθυμούμε να βελτιωθεί η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα. Αυτό σημειώνεται σε μεγάλο βαθμό. Σημείωσα την παρέμβαση του Προέδρου Σίση στο Κοινοβούλιο, όπου έγινε λόγος για πραγματικές πολιτικές εξελίξεις, για μεγαλύτερη ανεκτικότητα και δημιουργία κοινών χώρων. Τι πιστεύετε, μπορεί να γίνει μια, υπο, μια επίσκεψη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αίγυπτο για να ε, συζητήσουμε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σας. Μπορεί να γίνει μια τέτοια επίσκεψη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, συνήθω εδώ κάνουμε το εξή. Ε, Ποβάλλονται όλε τι ερωτήσει και μετά εσεί έχετε την δυνατότητα να απαντήσετε. Για του σοσιαλδημοκράτε, ο κύριος Σολέ. Όχι, όχι. Ε, λάθος, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Καν. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θίξω το εξή. Μιλήσατε για τη Μέση Ανατολή και για πάρα πολλέ άλλε χώρε και είπατε μόνο μία λέξη για τη λωρίδα τη Γάζα. Και ρωτώ, η Αίγυπτος τι μπορεί να κάνει για την κρίση τη Μέση Ανατολή, πώ μπορεί να παίξει ρόλο. Αναφερθήκατε σε όλε τι χώρε, αλλά δεν αναφερθήκατε καθόλου στην ε, σύγκρουση που υπάρχει μεταξύ, στη σχέση, στην κατάσταση Ισραήλ και λωρίδα τη Γάζα. Θέλω επίση να ρωτήσω το εξή. Αναφερθήκατε σε διάφορου ε, νόμου, αλλά ξέρετε, εγώ είδα πρόσφατα ε, τις διαδηλώσεις ε, που υπήρξαν για να απελευθερηθεί ένα σημαίνον στέλεχος της αντιπολίτευσης. Εξακολουθεί να υπάρχουν πολλοί ε, πολιτικοί κρατούμενοι στην Αίγυπτο. Υπάρχει και το θέμα μιας Ιταλίδας που δολοφονήθηκε στην Αίγυπτο. Πώς προχωράει η έρευνα η έρευνα για τον Τζούλιο Ρετζάνη, πώς ακριβώς προχωράει και αυτή, θα ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καλωσορίζουμε τον πρόεδρο, τον δόκτορα Αμπτουλά, Αμπτέλα Λάλ. Ε, έχω πάει δύο φορές στην Αίγυπτο και νομίζω ότι πρέπει να αναπτυχθεί η Αίγυπτος. Θέλω να ρωτήσω για την τουριστική αστυνομία, γιατί είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια για τους ε, τουρίστες που μεταβαίνουν στη χώρα σας. Αυτή η τουριστική αστυνομία υπάρχει ακόμα. Ε, να μπορούν εκεί να απευθυνθούν οι τουρίστες. Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω εξή. Αναφερθήκατε πολύ προσεκτικά βέβαια στην ελευθεροτυπία και είπατε ότι είναι ένας βασικός πυλώνας ε, της νέας νομοθεσίας και του συντάγματος. Και ρωτώ, ισχύει αυτό και για τον ξένο τύπο, παρήματος χάρη για το κανάλι Al Jazeera. Εμείς είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελευθερία του τύπου. Είναι καθοριστικό στοιχείο της ε, δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω ε, και για τη διένεξή σας με το Κατάρ ε, πώς μπορείτε και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να λύσετε αυτή την διένεξη με το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι από τους φιλελεύθερους, λέει ο κύριος Και θα ήθελα να μιλήσω για το ότι ανησυχούμε για την καταστολή εκδηλώσεων της ε, κοινωνίας των πολιτών, κυρίως τον περασμένο μήνα. Έχουμε ανησυχία για μεμονωμένες περιπτώσεις, blogger, και επίσης και ανεξάρτητων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αμαλφατή, παραδείγματος χάρη, που ανήρτησε ένα βίντεο για σεξουαλική παρενόχληση και μετά από λίγους μήνες συνελήφθη. Ε, εμείς ανησυχούμε, όμως έχασαν, ε, αφέθηκε ελεύθερος ε, με εγγύηση ε, μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την περίπτωση ε, ξένων χορηγήσεων αλλά και την ολοκλήρωση που θα υπάρξει στη διαδικασία για τα πολύ δρακόντια μέτρα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών και ε, ξένες παρεμβάσεις. Θα ήθελα να παρέμβω και εγώ για, τον, για τη Μωσέ Χασάν, που είναι πολύ γνωστή ακτιβίστρια της Αιγύπτου. Εχθές ε, ανακρίθηκε από τον δικαστή και είναι μία από τους υπέρμαχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει να αντιμετωπίσει πολύ βαριές ε, κατηγορίες με βάση την διάταξη 173 του ποινικού δικαίου. Και ε, κατηγορείται για το ότι ζήτησε να απελευθερωθούν ε, πολύ σωστά γυναίκες κρατούμενες. Εσείς τι έχετε να πείτε σχετικά με, αυτήν την, με το ενδεχόμενο της απελευθέρωσης γυναικών ε, κρατουμένων. Το δικό σας το Κοινοβούλιο έχει επιληφθεί του θέματος αυτής και ενδεχομένως και άλλων παρεμφερών ε, περιπτώσεων. Ο κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το ότι ε, έχετε επιδείξει κάποια συνέπεια και επιμένετε ε, σε αυτό που λέει η χώρα σας για τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ευρώπη. Τρομοκρατία και μετανάστευση. Σας άκουσα να μιλάτε ως τέλοχος της Αφρικής, ξέχουσα προσωπικότητα για αυτά τα δύο θέματα, μιλήσατε ξεκάθαρα. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις πολιτικές που είναι προς το κοινό συμφέρον. Ε, το πρόγραμμα Marshall, ο πρόεδρος κύριο Ταγιάννη τοποθετήθηκε από αυτού, αλλά θα θέλαμε να καθυστερήσουμε τη συγκεκριμένη εφαρμογή, την εκταμείευση των κονδυλίων. Η χώρα σας πρέπει να στηριχθεί από την Ευρώπη. Πολύ σημαντικό είναι η ανάπτυξη του τουρισμού, γιατί σήμερα ε, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς οι τουρίστες που μεταβαίνουν στην ε, Αίγυπτο και πολύ σημαντικό είναι και το θέμα των επενδύσεων. Εκεί νομίζω θα έχετε την αμέριστη υποστήριξη της Ιταλικής κυβέρνησης. Ο κύριος Σουπχάτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις πολύ σαφές εξηγήσει για τον τρόπο με τον οποίο μεταλλάσσεται η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και κινείται προς την κατεύθυνση περισσότερων ελευθεριών πολιτικών και οικονομικών. Καταλαβαίνω ε, τις ανάγκες που έχει η Αίγυπτος για ύπαρξη καθεστώτος ασφαλείας γιατί αντιμετωπίζει τρομοκρατικές απειλές και οφείλει να παίρνει τα μέτρα της. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Ποια είναι η άποψή σας για το ενδεχόμενο να έχουμε κέντρα υποδοχής στις νότιες όχθες της Μεσογείου όπου θα γίνεται η επεξεργασία των αιτημάτων ασύλου. Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε ενώπιον μιας μεταναστευτικής ροής άνευ προηγουμένου και θα ήταν σημαντικό να μας βοηθήσει η Αίγυπτος να εξετάσουμε όλα αυτά τα αιτήματα. Μπορεί η Αίγυπτος να είναι ε, αξιόπιστος εταίρος για να έχουμε τέτοιου είδους κέντρα υποδοχής και επεξεργασίας αιτημάτων ε, ασύλου. Κύριος Επιτίδιος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής Αιγύπτου, σας καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω να σας απευθύνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι να μας ενημερώσετε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις σχέσεις της Αιγύπτου με την Τουρκία. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν γνωρίζετε εάν από πλευρά Αιγύπτου υπάρχει η διάθεση να οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας με εκείνη της Ελλάδος όταν αυτή ανακηρυχθεί με τρόπο που να περιλαμβάνει το τμήμα της Μεσογείου που βρίσκεται ανατολικά της Κρήτης μέχρι το Τριεθνές της Κύπρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μαντάμ Αλίου Η κυρία Αλίου παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά γιατί μιλήσατε στα γαλλικά στην παρέμβασή σας. Η Αίγυπτος είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, απαραίτητη για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Έχω τρία ερωτήματα να σας θέσω. Πρώτον, ποια είναι η θέση και ο ρόλος της Αιγύπτου και του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου σε σχέση με την επίλυση των διαφόρων κρίσεων τις οποίες αναφέρατε, συμπεριλαμβανομένες της κρίσης μεταξύ των χωρών του κόλπου. Ποιο ρόλο θέλετε να αναλάβετε εκεί. από εκεί και πέρα. Σε σχέση με την τρομοκρατία, μας υπενθυμίσατε διάφορες δράσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι πολύ γνωστή η ποιότητα της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών και στην Ευρώπη κάνουμε σημαντική δουλειά για την απορριζοσπαστικοποίηση των πιο ακραίων στοιχείων. Έχετε εμπειρία που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας για τα θέματα αυτά. Τρίτον, η ισορροπία μεταξύ των κοινοτήτων είναι πολύ σημαντική για τη σταθερότητα της Αιγύπτου. Σήμερα η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση έχει και κόπτες στις τάξεις της. Δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται αυτό και στο Σύνταγμα. Ευχαριστώ. Κύριε Λοχμπίλα, κύριε Πρόεδρε, και εγώ έχω μία ερώτηση που αφορά στον Τζούλιο Ρετζίνη. Το θίξατε, εφήγη προηγουμένως. Από το 2016 οι συνάδελφοι από το Κοινοβούλιο τη Αιγυπτού μας λένε ότι υπάρχουν προσπάθειες για να το αποδοθεί δικαιοσύνη. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε ε, μέχρι το τέλος αυτής της ε, θητεία της κυβέρνηση, τι σκοπεύετε να κάνετε για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για μα αν τελικά μας καλέσετε ω Επιτροπή, ως Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επισκεφτούμε την Αίγυπτο και να συζητήσουμε επιτόπου στο Κάιρο. Και κατόπιν υπάρχουν και περιπτώσεις ε, ανθρώπων ε, που συνελήφθησαν πρόσφατα. Η μητέρα του Τζούλιο Ρετζίνη έχει κατέβει σε απεργία πείνας. Χάιταμ, παραδείγματος χάρη, ε, είναι blogger, ακτιβιστής και αυτοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες διότι τους αποδίδεται η κατηγορία του τρομοκράτη. Κύριε Πρόεδρε, 11 συνάδελφοι έβαλαν, υπέβαλαν ερωτήσεις, άρα βλέπετε πόσο σημαντική είναι για μας ε, η Αίγυπτος. 11 είχαν 11 ε, λεπτά χρόνο να ρωτήσουν και εσείς όμως θα πρέπει να είσαστε σύντομος γιατί μετά θα έρθει ο Σέιχης από το Κατάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολλά ερωτήματα μου τέθηκαν. Μήπως το καθένα χρειάζεται μια ολόκληρη συνεδρίαση, εγώ αυτό νομίζω. Και όλες οι ερωτήσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Συνοπτικά λοιπόν μπορώ να σας πω τα εξής. Η επίσκεψη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αίγυπτο είναι επιθυμητή. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια στη Μεσόγειο, αλλά και στην Αίγυπτο, την ελευθερία του τύπου, τα προβλήματα με τους ε, υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα προβλήματα στην Ευρώπη τη Μέση Ανατολή, η κρίση στη Γάζα. Αλλά και ό,τι έχει να κάνει με τη βοήθεια προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Ιταλό συνάδελφο που πρότεινε ένα σχέδιο Μάρσαλ για την Αίγυπτο. Όντως, βασιζόμαστε σε εσά. για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο Μάρσαλ για τη χώρα μου. Ξεκινώ λοιπόν με το πρώτο ερώτημα. με την επίσκεψη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αίγυπτο. Θα είναι χαρά για μένα, ως πρόεδρος του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου, να υποδεχθώ την αντιπροσωπεία αυτή στην Αίγυπτο. Είμαστε πολύ ανοιχτοί, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Και αν οι φίλοι μου από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιθυμούν να επισκεφθούν την Αίγυπτο, εμείς, ε, για εμάς είναι απολύτως ευπρόσδεκτοι. Όποτε το επιθυμήσουν. για τον Τζούλιο Ρετζίνη. Πρέπει να πω ότι η Αίγυπτος και η Ιταλία έχουν πολύ στενή συνεργασία. Η εισαγγελική αρχή της Αιγύπτου και η εισαγγελική αρχή της Ιταλίας, οι Αρμόδια, συνεργάζονται στενά γίνεται δουλειά, υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές. για να φτάσουμε στην αλήθεια και στην πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης. Τα προβλήματα με τον νόμο αναφορικά με τον τύπο έχουν ως εξής. Ο νόμος αυτός ισχύει και εφαρμόζεται για κάθε είδους τύπου, για κάθε είδους μέσα μαζικής επικοινωνίας και για τον Αιγυπτιακό τύπο αλλά και για τον ξένο τύπο. Δεν υπάρχει ποινή φυλάκισης για παράδειγμα για αδικήματα που διαπράττει κάποιος που εργάζεται στον τύπο με αυτή την ιδιότητα, είτε το γραπτό τύπο, είτε τον, το τηλεοπτικό μέσο επικοινωνίας. Τώρα για το θέμα της Λωρίδας της Γάζας, η Αίγυπτος έχει προσπαθήσει να συγκεντρώσει και να συνενώσει τα Παλαιστινιακά κόμματα ή για παράδειγμα τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή να τη συνενώσει. Κατάφερε να μιλήσει και με τα δύο αυτά κόμματα και έχει καταφέρει να πετύχει συμφωνία μεταξύ των δύο αυτών μερών Δυστυχώς υπάρχουν άλλα ξένα κόμματα που προσπαθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να διαταράξουν αυτή την συμφωνία και να την ε, διακόψουν. Η Αίγυπτος αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες της όσον αφορά στους Παλαιστινίους που διαβιούν και κατοικούν στη λωρίδα της Γάζας την τελευταία εβδομάδα και τον τελευταίο μήνα έχει στείλει πολύ μεγάλη βοήθεια. Βοήθεια επισητιστική, διατροφική και υγειονομική. Τώρα για τις άλλες συγκρούσεις στην περιοχή, είτε στην Ιεμένη είτε στη Συρία, έχουμε να πούμε ότι η Αίγυπτος προσπαθεί με κάθε μέσο να επιτύχουμε μια ειρηνική διευθέτηση όλων αυτών των συγκρούσεων. Στην Αίγυπτο, εάν κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ένα αδίκημα, βεβαίως πρέπει να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Και το δικαιοδοτικό σύστημα στην Αίγυπτο απλώνεται σε τρεις βαθμίδες. Δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη παρά μόνο εάν έχει επιληφθεί του θέματος η δικαιοσύνη σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. Υπάρχει προσωρινή κράτηση, όπως είναι η περίπτωση εδώ, και έχει και ανώτατο όριο τρεις μήνες η προσωρινή αυτή κράτηση. Και πρέπει πριν παρέλθει αυτή η προθεσμία να ε, υπάρξει η δίκη. Εάν λοιπόν έχουμε σε αυτή τη στιγμή ε, ε, υπερμάχων των ανθρώπινων δικαιωμάτων π.χ. Αυτό είναι μια προσωρινή κράτηση και ποτέ δεν μπορεί να διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Άρα δεν πρέπει να μιλούμε για φυλάκιση ή παράνομη φυλάκιση των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επανέρχομαι στο θέμα της αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Ελπίζω και να έρθετε και να συμμετάσχουν και μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην αποστολή αυτή στην Αίγυπτο. Είστε απολύτως ευπρόσδεκτοι όποια ημέρα θα θέλατε. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταλλαγή απόψεων, για το ότι απαντήσατε σε πάρα πολλές από τις ε, ερωτήσεις μας. Ήσασταν απόλυτα σαφείς ότι η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ευπρόσδεκτη στην Αίγυπτο. Και επιτρέψτε μου να σας ε, πω και εκ μέρους της Επιτροπής μας ότι ευχόμαστε στην Αίγυπτο κάθε επιτυχία γιατί θέλουμε στην περιοχή μια ισχυρή και σταθερή χώρα και θεωρούμε ότι η δική σας χώρα είναι βασικός δικός μας μας εταίρος. Ας παραμείνουμε λοιπόν σε στενή συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Καλή διαμονή στις Βρυξέλλες και καλή επιστροφή στη χώρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. δεν ήξερα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 Ladies Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε λοιπόν τώρα τη συνεδρίασή μας. Είμαστε στο σημείο υπερθμών 18 και πρέπει να σας πω, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας να μπορούμε να καλωσορίσουμε την αυτοεξοχότητα των Σεήχη Μοχάμετ Πιν Αμπτουλουράμ Πιν Γιασί Μαλτάνη, από το Κατάρ, ο οποίος συνοδεύεται από πολλά στελέχη, από πολλά στελέχη της ε, κυβέρνησής του και ε, από τον γνωστό σε όλους μας ε, στέλεχος ε, της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ καλές σχέσεις με όλες τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου και του Κατάρ. Οι σχέση με το Κατάρ είναι πολύ σημαντικές για μας. Αυτή η σχέση πρόσφατα ενισχύθηκε γιατί υπογράφηκε και η Συμφωνία Συνεργασίας τον Μάρτιο του 2018. Και αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει σε βάθος διάλογος ουσιαστικά ουσιαστική συνεργασία σε διάφορους τομείς. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες διαφοροποίησης ε, του Κατάρ ε, με βάση ε, το όραμα του 2030. Εσείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε τοποθετηθεί με ουδέτερο τρόπο στην συνεχιζόμενη κρίση στον κόλπο και μετά από ένα χρόνιο, χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να έχει την ίδια σχέση. Εμείς θεωρούμε ότι η συνοχή είναι καθοριστική σημασία σημασίας για την ε, περιοχή, για τη σταθερότητα τη περιοχή. Όλοι μα ε, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τι τελευταίε εξελίξει. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τι τελευταίε εβδομάδε. Πιστεύουμε ότι η αποκλιμάκωση είναι καθοριστική σημασία για να επιτευχθεί η περιφερειακή σταθερότητα. Η κρίση θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε ε, να βγει κανεί πιο ενδυναμωμένο από αυτή την κρίση. Και αυτό είναι το μήνυμα που ε, στείλαμε πριν από μερικούς μήνες όταν επισκεφτήκαμε το Ριάντ ε, Εξοχότατε, σας καλέσαμε γιατί θέλουμε να μας ενημερώσετε για τις απόψεις του Κατάρ για την κρίση του κόλπου, το πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα και κατά πόσον συμμερίζεστε τις ε, απόψεις Αμερικής ότι θα πρέπει να γίνει ε, μια ναι, εκ νέου συνάντηση, το Camp David, αυτή έχει τώρα αναβληθεί για το Σεπτέμβρη. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Ε, σας καλωσορίζουμε θερμά. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που μου δίνουν σήμερα την ευκαιρία να τους απευθύνω το λόγο. Με φιλοξενείτε, έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ σε εσά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την εξωτερική πολιτική του Κατάρ και με την εσωτερική πολιτική επίσης και πώς ακριβώς έχει ε, επιβιώσει σε αυτή την ε, δύσκολη περίοδο, κυρίως στις αναταραχές ε, οι οποίες μας ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η κοινωνική και η οικονομική ανάπτυξη βρίσκεται στην καρδιά της ανάπτυξης του Κατάρ και αυτό πρέπει να πω, δεν αφορά μόνο την εσωτερική πολιτική, αλλά αυτές είναι και οι αρχές που διέπουν την εξωτερική μας πολιτική. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε προβεί σε πολύ μεγάλες επενδύσεις, έτσι ώστε να προάγουμε αυτές τις αξίες που πρεσβεύουμε στη Μέση Ανατολή. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, εμείς έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το Κατάρ έχει επενδύσει έχει προβεί σε μεγάλες επενδύσεις στην εκπαίδευση. Τώρα είναι γνωστό το Κατάρ για πανεπιστήμια υψηλού κύρους, ε, επίσης ε, και για τα σχολεία μας, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της ακαδημαϊκής έρευνας στη χώρα μας. Αυτό είναι μοναδικό στην περιοχή. Και επίσης, ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκεί έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Πλέον έχουμε κανόνες, κανονισμούς για να προστατεύονται οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργατικών δικαιωμάτων και για να αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στη διεθνή κοινότητα. Η βελτίωση της θέσης των γυναικών. Αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες της εσωτερικής πολιτικής του Κατάρ και μάλιστα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των ε, γυναικών στην ε, δική μας τη χώρα. Οι γυναίκες ε, είναι ποσοστιαία πολύ περισσότερες από τους άρενες στην, σε επίπεδο εκπαίδευσης. Όσον αφορά την στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε επενδύσει τα τελευταία 20 χρόνια ε, ουσιαστικά στο να προσφέρουμε μία πλατφόρμα για ένα διάλογο ανάμεσα στις ομολογίες και τα δόγματα. Κατά τα άλλα, έχουμε επίσης εστιάσει την προσοχή μας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, γιατί πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα επέλθει ευημερία στους πολίτες μας. Θα ελέγχουμε βέβαια την, και την ελέγχουμε την πρόοδο ε, του Κατάρ τα τελευταία 10 χρόνια και καταλήξαμε στο ότι σήμερα το Κατάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ενέργειας στην παγκόσμια αγορά. Το 30% του υγροποιημένου αερίου στον κόσμο προέρχεται από το Κατάρ. Άρα δηλαδή Μιλάμε για ένα καθοριστική σημασία εταίρο για πάρα πολλές χώρες και ευρωπαϊκές ε, και την Ασία. Και η Ευρώπη όμως να επανέλθω είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για μας μετά την Ασία, ενώ η Ιαπωνία και Κορέα. Το υγροποιημένο αέριο το προμηθεύουμε στην Πολωνία, στον Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το Κατάρ λοιπόν έχει αποδείξει τις τελευταίες δύο δεκαετίες ότι είναι ένας αξιόπιστος εταίρος σε θέματα ενέργειας. Επίσης, αν δείτε λιγάκι το μέγεθος της οικονομίας μας και ε, στρέψτε το βλέμμα στο 98 ε, το ΑΕΠ μας ήταν περίπου 10 δις δολάρια. Σήμερα ξεπερνάμε τα 150 δις δολάρια, που σημαίνει 15 ε, φορές έχει αυξηθεί το ΑΕΠ μας μόνο μέσα σε δύο δεκαετίες. Αυτή λοιπόν η ανάπτυξη και η πρόοδος κατ' ήταν το αποτέλεσμα πολλών προσπαθειών που ανέλαβε η κυβέρνηση αλλά και ο λαός του Κατάρ. Και αυτά συμβάλλουν στην ευημερία όχι μόνο της ε, χώρας μας αλλά επίσης και στην ευημερία της ευρύτερης περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για μας. Το 30% ε, των εισαγωγών μας, αναφέρομαι τώρα στις εισαγωγές, προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κατάρ τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει επενδύσει ουσιαστικά στην ελευθερία πρόσβασης στην ενημέρωση και στα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Πράγματι είμαστε μια περιοχή όπου τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι τόσο ελεύθερα όπως εδώ, στη Δύση, αλλά εμείς, εν πάση περιπτώσει, είμαστε καλύτεροι από τους υπόλοιπους στην περιοχή, προσφέρουμε ελευθερία έκφρασης και όχι μόνο αυτό, αλλά καθορίζουμε και τα κριτήρια για τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Παραδείγματος χάρη, πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχαν ε, καθόλου ε, κανάλια ενημέρωσης ή πλατφόρμες ενημέρωσης για τον αραβικό κόσμο, εκτός από τις επίσημες ε, πλατφόρμες και τις κυβερνήσεις. Ε, το Κατάρ λοιπόν έχει και στηρίξει και χρηματοδοτήσει την ίδρυση του Al Jazeera, που τώρα πλέον είναι ένα κανάλι ενημέρωση παγκοσμίου εμβέλεια και αναγνώριση, όχι μόνο στα αραβικά, αλλά και στα αγγλικά και σε άλλε γλώσσε. Επίση, πιστεύουμε ότι ο επικοδομητικός διάλογος είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός για να υπάρχει συνύπαρξη και συμβίωση. Ε, το Κατάρ προσφέρει μια πλατφόρμα έτσι ώστε αντιμαχόμενες πλευρές να μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, ε, να προσπαθήσουν να ε, λύσουν τα προβλήματά τους μέσα από τον διάλογο και όχι τη σύγκρουση. Επίσης, η χώρα μας έχει επενδύσει τα μάλα στην ε, καλή διακυβέρνηση. Το κράτος δικαίου ε, είναι σεβαστό στο Κατάρ, ιδιαίτερα σεβαστό μάλιστα, και είμαστε πεπισμένοι ότι η διαφάνεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα από τα καθαριστικά στοιχεία για την ε, επιτυχία της χώρας μας. Το Κατάρ λοιπόν έχει αποδείξει ότι είναι πρωτοπόρα χώρα τα θέματα αυτά στην περιοχή. Και μάλιστα το Κατάρ είναι το πρώτο στην ε, κλίμακα ε, εμπιστοσύνης ε, των υπολείπων για τη λήψη αποφάσεων και σε σχέση και με την αποτελεσματικότητα του, των νόμων και της νομοθεσίας. Υπάρχουν λοιπόν για μας αυτές οι αρχές και οι αξίες οι οποίες αποτελούν τη βάση, τα θεμέλια της περιοχής. Εμείς όλα αυτά τα ενστερνιζόμαστε, προσπαθούμε να τα διαδώσουμε περαιτέρω, αξίες δηλαδή τις οποίες καταρχήν έχουμε ενστερνιστεί και μετά προσπαθούμε να τις ε, διαδώσουμε. Το θέμα είναι δηλαδή πρώτα να υιοθετούμε και να εφαρμόζουμε κάποιες αξίες και μετά να προσπαθούμε να πείσουμε άλλες χώρες του κόλπου να αγκαλιάσουν και αυτές, αυτές τις αξίες. Εμείς ε, αυτό, όπως σας είπα, το έχουμε πράξει προσφέροντας κυρίως ε, την ε, βοήθειά μας ε, σε άλλες αδελφές χώρες της Μέσης Ανατολής. Παράδειγμα της διαβούλευσης και των, της διαμεσολάβησης που έχουμε προσφέρει σε 10 συμφωνίες ειρήνης, εκεί είτε έχουμε διαμεσολαβήσει είτε έχουμε στηρίξει συμφωνίες με το Λίβανο, το Σουδάν, συμφωνία ανάμεσα συμφωνία με τους Παλαιστίνιους. Επίσης, έχουμε προσφέρει πολλές ευκαιρίες έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τον Απρίλιο εγκαινιάσαμε προγράμματα που στήριζονται κυρίως από το Κατάρ, από την κυβέρνηση του Κατάρ. Συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και της Ευρώπης και πλέον έχουμε 10 εκατομμύρια παιδιά τα οποία έχουν αποφυτίσει. Και αυτό το γεγονός το εορτάζουμε. Η οικονομική ανάπτυξη είναι η βασική κινητήρια δύναμη για την ευημερία. Εμεί έχουμε προβεί σε επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στο Κατάρ. Έχουμε πλέον θεσμού που προσφέρουν πάρα πολλέ ευκαιρίες σε εκατοντάδες ε, χιλιάδες ε, νέους ε, στην περιοχή μας. Επίσης, το να προσφέρει κανείς ε, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ε, σε πολίτες, κυρίως σε ευάλωτες ε, κοινωνίες, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επικρατήσει περαιτέρω σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό εμείς έχουμε στηρίξει προγράμματα νοικοδόμησης στο Λίβανο, στο Νταρφούρ, στο Σουδάν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο Σουδάν οι εκτοπισμένοι του Νταρφούρ τώρα πλέον αρχίζουν να επανέρχονται στις γενέτηρές τους. Γιατί εκεί έχουν τη δυνατότητα σχολικής εκπαίδευσης, ε, κατοικίας, ε, κέντρα υγείας. Όλα αυτά λοιπόν ε, αποτελούν ένα τμήμα του οράματος του Κατάρ για την περιοχή. Νομίζω εσείς ως μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί κυρίως η Εμένη, η Σομαλία, η Λιβύη, η Συρία, η διεθνικός, διασυνοριακό ε, ε, και τρομοκρατία και η πρόσφατη κρίση βλέπουμε ότι τελικά υπάρχει μια διασύνδεση στην κρίση της Μέσης Ανατολής και πιστεύουμε ότι η Μέση Ανατολή ε, πρέπει να στηρίξει την νοτροπία αυτή της ε, ασφάλειας ε, χωρίς αποκλεισμούς στη δική μας την περιοχή. Για να είμαστε λοιπόν ενωμένοι οι δυνάμεις της ε, περιοχής ε, επιδιώκουν την ε, περισσότερη σταθερότητα και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Στα πολιτικά. Γίνονται χειρισμοί στην Μέση Ανατολή. Υπάρχουν μη επικοδομητικά μέτρα. Αυτά βλάπτουν την ασφάλεια προκύπτει ένα κενό εξουσίας και αυτό το κενό κατ' ουσίαν αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για την τρομοκρατία και το ριζοσπαστισμό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίστακτη συμπεριφορά και η δική μου η χώρα και αυτή η πέστη ε, τη από κάποιες από αυτές τις ε, πολιτικές ε, μέσα σε μια νύχτα οι γείτονές μας λένε ότι οι αλλαγές που έχουν επιφέρει κάποιοι άλλοι, αυτό είναι απειλή. Και όποιος ε, διαφωνεί, ε, ονοματίζεται τρομοκράτης. Εμείς ε, στο Κατάρ δεχόμαστε την επικοδομητική κριτική για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις χώρες μας. Βλέπουμε όμως επίσης ότι η συμφωνία, το αποτέλεσμα σε αυτή τη συμφωνία δεν είναι ο αποκλεισμός. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση, εμείς ζητήσαμε από τους γειτονές μας να συναντηθούμε σε τράπεζα διαπραγματεύσεων, να συζητήσουμε, να εξηγηθεί το θέμα του αποκλεισμού Υπάρχει αυτό το, η μοναδική ε, μορφή και ο χαρακτήρας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, αλλά δυστυχώς ε, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση κλιμακώνεται περαιτέρω από τους γείτονές μας. Οι γείτονές μας αγνοούν την πορεία που έχει χαράξει η διεθνής κοινότητα αρνούνται το διάλογο και προτείνουν ε, μη επικοδομητικά μέτρα και έναντι άλλων χωρών της περιοχής. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η δική μας περιοχή δεν μπορεί να δεχτεί και άλλη κρίση. Ήδη υπάρχουν αρκετές κρίσεις. Υπάρχουν αρκετές αρνητικές ε, επιπτώσεις στη χώρα μας, στη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλες οι χώρες μέση Ανατολής να εμπλακούν στην ε, περιφερειακή σταθερότητα. Γιατί παντού ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, οι ίδιοι πρωταγωνιστές, αυτοί είναι που θα πρέπει να έρθουν στην τράπεζα διαπραγματεύσεων και με βασικό μέλημα την ασφάλεια να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί οτιδήποτε πάει στραβά στη δική μας περιοχή θα μετακυλιστεί, θα διαχυθεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα υπάρχουν περισσότεροι μετανάστες, ε, θα οξυνθεί η κρίση, ε, θα έχουμε πιο έντονη τη διεθνή τρομοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, χαιρετίζουμε την προσπάθεια των ευρωπαϊκών κρατών να στηρίξουν τον διάλογο για την σταθερότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Your Σας ευχαριστώ πολύ, εξοχότητα. 20 λεπτά έχουμε περίπου για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Προς στιγμή έχω πέντε συναδέλφους οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Λοχπίλα Πέντε λοιπόν ομιλητές, αλλά πριν θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Λιωμαρή που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας με τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ε, Υπουργέ, ε, εξοχότης, θα ήθελα να σας καλωσορίσω πρώτα απ' όλα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ας περιμένουμε λίγο να βάλετε τα ακουστικά σας. Θα μπορούσα να μιλήσω και αγγλικά, λέει η κυρία Λιωμαρία, αλλά καλύτερα είναι και για σας και για μένα να μιλήσω γαλλικά. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύντομα θα τα πω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, μας πιέζει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να θέσω τρία ερωτήματα. Το Κατάρ παίζει οικονομικό αλλά και πολιτικό ρόλο ουσιώδη ε, σε μια στρατηγική σημασία περιφέρεια ε, και για την ανάπτυξη αλλά και για την ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής και της Ευρώπης ε, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Ξεκινώντα από αυτή τη σκέψη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή Σε οικονομικό επίπεδο, ποιοι είναι οι κατά προτεραιότητα τομείς οικονομικής διαφοροποίησης της χώρας σας. Ε, διαφοροποίηση οικονομική για το ίδιο το Κατάρ, αλλά και εκτός του ε, Κατάρ μέσω των επενδύσεων που κάνετε. Ποιοι είναι οι τομείς που επιλέγετε και ποιες είναι οι γεωγραφικές περιφέρειες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Δεύτερη ερώτηση ε, που αφορά την πολιτική και τη στρατηγική είναι ε, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Θα μπορούσατε να μας πείτε, δίνοντας κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, ποια είναι τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιεί το Κατάρ για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία. Ε, δηλαδή είτε πρόκειται για ε, την απορριζοσπαστικοποίηση είτε πρόκειται ε, για την, τον έλεγχο των χρηματικών ροών. Τρίτο στοιχείο της κρίσης που αναφέρατε όσον αφορά το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, θεωρείτε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα του επόμενου μήνε. Έχουμε την αίσθηση μερικέ φορέ ότι κινούνται λίγο τα πράγματα, αλλά άλλε φορέ έχουμε την αίσθηση ότι αυτή η κρίση θα κρατήσει χρόνια. Ε, έγινε μια συνεδρίαση ε, του Συμβουλίου στο Κουβέιτ, αλλά ήταν τεχνικού χαρακτήρα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια για πολιτικές επαφέ του επόμενου μήνε, τα επόμενα χρόνια. Τελευταία ερώτηση. Αναφερθήκατε στι αξίε και τι μεγάλε αρχέ που εφαρμόζει το Κατάρ. Δύο ερωτήματα μας απασχολούν εδώ. Πρώτον, ε, το πρόβλημα της ε, θρησκευτικής ε, ανεκτικότητας. Αν έχετε πάρει κάποιες, αναλάβει κάποιες προτεραιότητες. Και δεύτερον, το θέμα των ξένων εργαζομένων. Γιατί ξέρετε ότι και για αυτό το θέμα έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λιωμαρή, λέει ο Πρόεδρο και δίνω λοιπόν το λόγο τώρα στου άλλου συναδέλφου. Προτείνω, ε, ε, να ε, απαντήσετε συνολικά στι ερωτήσει. Εν τω μεταξύ όμως έχουν εγγραφεί οκτώ ομιλητές. Ένα λεπτό ο καθένας θα έχετε. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ο κύριος Αλαφράγκα πρώτος. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Πριν από ένα χρόνο ε, ε, διακόπησαν οι διπλωματικές ε, σχέσεις της χώρας σας με τα Εμμυράτα, αλλά φαίνεται ότι δεν καταφέρατε να συνεχίσετε, δεν σήμανε ότι δεν είχατε πλέον διπλωματικές σχέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει το κόστος αυτής της κατάστασης είναι ότι χάνουν όλοι και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου χάνει και εσείς γιατί χάνετε οικονομικά, έχετε βεβαίω ε, αντοχέ ακόμα, αλλά κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε ποιε είναι οι προσδοκίε σα. Εμείς ε, πριν από λίγο καιρό σε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, ε, επισκεφθήκαμε το ε, Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία. Είχαμε εδώ επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικό του Ιράν. Πιστεύετε ότι μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη στην διαμεσολάβηση του Κουβέιτ των Ηνωμένων Πολιτειών και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση που είναι κακή για όλους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν καταγράφονται άλλοι ομιλητέ Έκλεισε ο κατάλογος. Ο κύριος Παντζέρη, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Εγώ ε, πολύ ε, σύντομα ε, θα αναφερθώ στην κρίση του κόλπου γιατί μας απασχολεί πολύ και μας ενδιαφέρουν πολύ οι εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να δεσμευτούμε έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι καλές προϋποθέσεις. Όπως έλεγε προηγουμένως και ο πρόεδρος Μακάλιστερ, η Ευρώπη θέλει να βοηθήσει, υποβοηθήσει τη διαμεσολάβηση του Κουβέιτ, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια επιπλέον βήματα. Ο καθένα θα πρέπει να κάνει ε, επιπλέον ε, βήματα. Το Κατάρ για να καταπολεμήσει περισσότερο την τομοκρατία ε, και να συνεχίσει στην οδό της διεύρυνσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την πλευρά τη Ευρώπη, όμως θα πρέπει επίσης να γίνει δουλειά. Θα πρέπει να διευκολύνει το διάλογο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσει ισορροπημένη θέση. Πιστεύω ότι καλή ιδέα θα ήταν, α πούμε, εάν η ίδια η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για τη σχέση με την Αναβική Χερσόνησο έπαιρνε μια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μπασίρ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ε, αξιοχώτης, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Χαιρετίζω τις προσπάθειες που καταγράφει η χώρα σας ε, για το Jazeera, για μια αντικειμενική πλατφόρμα. Έχω δύο ερωτήσεις για σας. Πρώτον, θα ήθελα να σχολιάσετε ε, ε, την, το, να σχολιάσετε την θέση των πολιτών σας σε σχέση με την, τον αποκλεισμό δηλαδή δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών κτλ. Επίσης ε, θα θέλατε ε, εν τέλει κάποια διαμεσολάβηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από το Κουβέιτ και το Ομάν. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Λέει η κυρία Βαλίνα Ντελανόβαλ. Θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε με το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για δύο κράτη Ισραήλ-Παλαιστίνης. και την άποψή σας για τις τελευταίες, ε, τις πρόσφατες εξελίξεις και την βία στην ε, ε, Γάζα. Όσον αφορά την τρομοκρατία και την καταπολέμησή της, πιστεύετε ε, ότι τέτοιου είδους πολιτικές, ε, δηλαδή τον εξωθεί κανείς τον κόσμο στην απελπισία, μια τέτοια απάνθρωπη στάση όπως αυτή του Ισραήλ, πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή αντιθέτως πιέζεται ο κόσμος, εξωθείται να πάρει θέσεις τις οποίες δεν θα έπαιρνε διαφορετικά. Η κυρία Λόχ Μπίλερ για τους πράσινους, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις δηλώσει σας ε, κύριε Υπουργέ. Μία ερώτηση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κυρίω όσον αφορά τους μετανάστες εργαζόμενους. Πριν από χρόνια ε, κάναμε πολλές ακροάσεις ε, στο Κοινοβούλιο και είναι ενθαρρυντικό βέβαια που εσείς έχετε προωθήσει κάποιους πολύ προοδευτικούς νόμους όσον αφορά την προστασία των εργασιακών ε, ε, δικαιωμάτων. Αυτό ε, σας είναι πάρα πολύ θετικό. Υπάρχουν όμως κάποια νέα όσον αφορά και το την ελάχιστη αμοιβή. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Επίσης, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε και δύο λόγια όσον αφορά την ιεμένη αυτήν την σύγκρουση με τόσα, τόσες απάνθρωπες καταστάσεις και τόσα θύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική του Κατάρ ήταν εξαιρετικά αρνητική στην Συρία. Ε, και ε, χώρισε λίγο μετά από την διεθνή κατακραυγή. Ε, ξέρουμε ότι έχει βοηθήσει ομάδες όπως η Ασνούρα και άλλες το Κατάρα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η σημερινή άποψη του Κατάρα. Μάθατε από τα διδάγματα του παρελθόντος, μάθατε μετά από τον πόλεμο ότι δεν πρέπει να υποστηρίζετε ακραίες τρομοκρατικές ομάδες και επίσης ε, ποια είναι η θέση όσον αφορά το ε, Ιράν και την ε, διαρκώς πιο επιθετική πολιτική της Σαουδικής Αραβίας. Ευχαριστώ πολύ. Από τους μη γραμμένους ο Κάβερ. Um, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. μιλήσατε για διάλογο ε, υπάρχει δυνατότητα διαλόγου μεταξύ Κατάρ και Σαουδικής Αραβίας, επίσης ε, μεταξύ Κατάρ και Ιράν. Πιστεύετε ότι ε, υπάρχει καμία δυνατότητα να ασκήσετε πίεση έτσι ώστε να σταματήσει η ροή όπλων το Ιράν στην Ιεμένη. Και επίσης μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας μακροπρόθεσμα για την εξέλιξη στην Ιεμένη. επόμενη ομιλήτρια Ραμόνα Μανέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριε Υπουργέ. Ευελπιστώ ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με πιο ε, ε, έντονο ε, τρόπο. Εμείς να σας πω ότι έχουμε υπογράψει και συμφωνία με την Επιτροπή, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμπεριλαμβάνεται στις αναφορές μας και το Κατάρ. Είναι σημαντικό βεβαίως να σταθεροποιηθεί η περιοχή. Και όταν λέω ότι εμεί θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η περιοχή, αναφέρομαι βεβαίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό τη, από τη δικιά σα πλευρά. Έχετε σκεφτεί περαιτέρω συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουμε κοινά ε, συμφέροντα όσον αφορά την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας. Καθώς επίσης και όσον αφορά την ε, βοήθεια γενικότερα. Ο κύριος Καν. Ε, σε σχέση με τη διαμάχη με την Σαουδική Αραβία. Βεβαίως δεν είναι ε, κανείς ε, καλό να παρισφρεί σε κάτι το οποίο θα πρέπει να λύσει το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Αλλά όπως είπε και η κυρία Λιωμαρή προηγουμένως, ε, ε, ε, ίσως θα πρέπει να δούμε εάν μπορεί να προωθηθεί λίγο περισσότερο το θέμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δούμε ότι το, η διαμεσολεύση του Κουβέιτ δεν αρκεί. μιλήσατε για μεταρρυθμίσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι η ε, οι γυναίκες κυρίως που δουλεύουν ε, ως εσωτερικές βοηθοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργασιακή μεταρρύθμιση. Ε, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δέκα ομιλητές, αλλά τριάντα ήταν οι ερωτήσεις. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέει ο Πρόεδρος. Εάν κάποια δεν καταφέρω να την απαντήσω, παρακαλώ να μου το θυμίσετε. Και θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και συνοπτικός στα λεγόμενά μου. Όσον αφορά στην ερώτηση για τον οικονομικό και πολιτικό ρόλο του Κατάρ στο διεθνές στερέωμα. Μέρος του εθνικού μου ασοράματος είναι να προχωρήσουμε στην διαφοροποίηση της οικονομίας μας. Η πλειονότητα ε, του ΑΕΠ προέρχεται από τον τομέα των ανθράκων και θέλουμε να υιοθετήσουμε, έξω και το πράξαμε, το όραμα της διαφοροποίησης της παραγωγικής μας βάσης και γι' αυτό έχουμε σημειώσει πολύ καλή πρόοδο. Το 86% του ΑΕΠ ήταν, προερχόταν από τους υδρογονάνθρακες και το 2017 ε, είχε πέσει η συνεισφορά αυτή στο ΑΕΠ των υδρογονανθράκων στο 50%. Χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Επενδύουμε σε διάφορους κλάδους της οικονομίας Προσπαθούμε να αναπτύξουμε ε, κλάδους που να έχουν ε, ροή πιο ε, downstream και να καλύψουμε τις υποδομές αερολιμένων, λιμένων. Το Σεπτέμβριο επενδύσαμε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το λιμάνι του Κατάρ και τώρα ήδη έχει φτάσει στο 27% του διεθνούς αμπορίου που περνάει από αυτό τον λιμένα. Και όλα αυτά τα πράξαμε από νωρί, όταν η τιμή του πετρελαίου ήταν ψηλά. Αποφασίσαμε λοιπόν να επενδύσουμε το πλεόνασμα από τις πωλήσει πετρελαϊκών προϊόντων ε, και στο εξωτερικό. Κάναμε διεθνείς επενδύσεις και επιδιώξαμε να επενδύσουμε σε ε, εταιρείε περιοπής παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη, στην Ασία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως, βασικός αποδέκτης των επενδύσεών μας είναι η Ευρώπη. Είτε πρόκειται για το χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε για άλλους κλάδους της οικονομίας. Και οι επενδύσεις αυτές ε, πηγαίνουν αρκετά καλά. Αυτά λοιπόν για τη διαφοροποίηση της οικονομίας. Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας, Κάνουμε το παν για να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό στην περιοχή μας. Έχουμε διεθνή αναπτυξιακή ατζέντα, την οποία ανέφερα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Και μεγάλο μέρος αυτής την έχουμε αφιερώσει, το έχουμε αφιερώσει στην καταπολέμηση των βασικών αιτιών που προκαλούν την τρομοκρατία. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να εξεταστεί και από πλευράς επιχειρησιακής και από πλευράς στρατηγικής. Είμαστε στο επίκεντρο της συμμαχίας κατά του ΝΤΑΕΣ και στη δική μας επικράτεια υποδεχόμαστε τις δυνάμεις αυτού της συμμαχίας και οι ένοπλες δυνάμεις μας συμμετέχουν και προσφέρουν υπηρεσίες στήριξης και επιμελητίας. Επίσης ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και παρακολουθούμε στενά τα συστήματα αυτά που έχουμε. Το 2014 αρχίζαμε να ελέγχουμε τους εράνους που γίνονται από φιλανθρωπικές οργανώσεις, γιατί εκεί είναι ένας διάβλος που μπορεί να διοχετεύσει τα χρήματα σε λάθος χέρια. Έχουμε λοιπόν αναπτύξει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και έχουμε ασκήσει και διώξεις Συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε κάνει πολλά, αυτό είναι αληθές, αλλά μένουν και άλλα που πρέπει να γίνουν. Πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Άλλωστε, δεν είναι φαινόμενο που είναι καινούριο μόνο για μας, είναι κάτι το καινοφανές για τον υπόλοιπο κόσμο, για όλον τον κόσμο. Άρα οφείλουμε να συνεργαστούμε, να ενισχύσουμε το διάλογο και τη συνεργασία με διάφορες χώρες. Έχουμε υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες, η οποία προβλέπει τεχνική στήριξη και βοήθεια για την οικοδόμηση και τη δημιουργία δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Έχουμε υπογράψει σχετική συμφωνία με τη Γαλλία επίσης και έγινε ο πρώτος διάλογος για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πέρσι με τη Γαλλία για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και το συζητούμε και με άλλες χώρες και προσπαθούμε να ενισχύσουμε το δίκτυο ε, πληροφοριών που έχουμε έτσι ώστε να εντοπίσουμε καλύτερα τις πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θέλουμε να θωρακίσουμε το νομοθετικό μας πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση ακόμα περισσότερο. Από εκεί και πέρα. Μιλήσατε για την εχώρια μας πολιτική, για την πολιτική θρησκευτική ανεκτικότητας και ε, για τα δικαιώματα. Έχουμε επιβάλει διαθρησκιακό διάλογο τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι κάτι που το κάνουμε 20 χρόνια τώρα και πραγματικά το εφαρμόζουμε. Άνθρωποι από διαφορετικές θρησκείες μπορούν να ασκούν ε, θρησκευτικά τους καθήκοντα, να εκφράζουν τη θρησκεία τους ελευθέρως και έχουμε και χώρους λατρείας των χριστιανών που υπάρχουν και είναι διαθέσιμοι χώροι. Αυτή είναι σαφή σε εκδήλωση θρησκευτικής ανεκτικότητας. Σε άλλες χώρες κατάσχουν τους σταυρούς στα αεροδρόμια. Στο Κατάρ εμείς πιστεύουμε ότι για να έχουμε αρμονική συνύπαρξη είναι απαραίτητος αυτός ο διάλογος για να συμβάλλουμε θετικά στην πορεία της ανθρωπότητας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα, Πολύ μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Και εδώ έγκυται η εξή ειδοποιώ διαφορά. Μιλούμε για χώρα που δέχεται τις επικρίσεις και προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει επικοδομητικά και μιλούμε και για χώρες που δεν δέχονται καμία επίκριση και δεν επιτρέπουν και σε κανέναν να τους επικρίνει και λαμβάνουν μέτρα εναντίον οποιοδήποτε ασκεί, οποιοδήποτε είδους κριτική. Εμείς καλωσορίζουμε την κριτική. Έχουμε μέλη του δικού σας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν έρθει, μας έχουν επισκεφθεί τρία-τέσσερα χρόνια τώρα και μπορούν να δουν ότι έχουν σημειωθεί πολύ σημαντικές αλλαγές. Έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία και το διάλογο. Και χάρη στους φίλους μας. Έχουμε υπογράψει η συμφωνία μεταξύ της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της δικής σας και της δικής μας Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλουμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, με άλλους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης. Σημεριζόμαστε τις αξίες αυτές συμμεριζόμαστε τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν δεχόμαστε κάποιος να βρει το θάνατο στο χώρο εργασίας του γιατί ο εργολάβος ή ο κατασκευαστής δεν έχει τηρήσει την εργασιακή νομοθεσία. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά ε, αποτελέσματα για τους εργαζομένους, ε, για τους χειρονάκτες εργάτες και να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στις καλύτερες δυνατές συνθήκες συμβάλλουν ιδιαίτερο στην πρόοδό μας. Είμαστε μικρή χώρα και μικρός είναι ο μας και εκτιμούμε ιδιαίτερο σε αυτή την προσπάθεια. Επομένως έχουμε κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους εργαζομένων στα εργοτάξια, Πρέπει να πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη ένας θάνατος εργαζομένου ισοδυναμεί με όσα να είχαν βρει το θάνατο χίλι. Δηλαδή ο θάνατος ενός είναι εξίσου σημαντικός. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει ανεκτό. Ενισχύσαμε λοιπόν τους κανόνες, τους περιορισμούς, Εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας, έχουμε διπλασιάσει τις επιθεωρήσεις και τις εποπτείες, τον αριθμό των επιθεωρητών. Έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας. Έχει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ο ILO, τοπικά γραφεία στην Τόχα του Κατάρ και βοηθά το δικό μας Υπουργείο Εργασίας για να αποκτήσει τις κατάλληλες ε, δυνατότητες για να σημειωθεί πρόοδος και προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, κοιτάζοντας τις σημειώσεις μου, ε, προσπαθώ να τα απαντήσω όλα. Ερχόμενος λοιπόν στα περιφερειακά ζητήματα, για να σας πω για τις χορηγίες και το sponsorship, έχουμε νέα νομοθεσία και όλες οι εταιρείες αλλάζουν όπου οι συμβατικές σχέσεις και οι εργοδοτικές σχέσεις δεν ακολουθούν το σύστημα του sponsorship πια και τα αποτελέσματα είναι θετικά. Δύο λόγια για την κρίση στο κόλπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προχωρήσουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή το Κατάρ είναι ανοιχτό προς το διάλογο. Έχουμε εκφράσει την απόψή μας, ότι είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε διάλογο. Έχουμε ακούσει τις απόψεις και του Κουβέιτ, που είναι ο βασικός διαμεσολαβητής και θέλουμε οι διεθνείς εταίροι να στηρίξουν και τον Εμμύρη του Κουβέιτ. Εμείς έχουμε εμπλακεί σε συζήτηση Πρόσφατα, ο Εμμύρης του Κουβέιτ απέστειλε επιστολή προς όλες τις χώρες που είναι μέλη του Gulf Cooperation Council, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και το Κατάρ, ήταν η μόνη χώρα που απάντησε και θετικά μάλιστα στον Εμμύρη του Κουβέιτ. Στείλαμε την απάντησή μας πριν από τρεις εβδομάδες και καμία άλλη ε, χώρα δεν έχει ακόμα απαντήσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε επικοδομητική στάση και ότι η λύση θα βρεθεί μέσα από το διεύλο του ειρηνικού διαλόγου. Πιστεύουμε ότι όλοι χάνουν λόγω αυτής της κρίσης. Οι άνθρωποι μας χάνουν, ε, υπονομεύεται η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά χάνουν και οι διεθνείς ε, εταίροι. Και οι χώρες που μας έχουν επιβάλει αυτό το εμπάρκο προσπαθούν να αγνοήσουν το γεγονός ότι τελικά υπονομεύουν και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής. Τώρα, ως προς το μέλλον του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ελπίζουμε αυτό να είναι ε, με ευημερία και καρποφόρα, καρποφόρο, αλλά θα δούμε ποιες είναι οι δεσμευτικές αρχές ε, που επιβάλλουν στις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το Συμβούλιο να μην ε, κάνουν επίθεση σε αέτερο μέλος του Συμβουλίου θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι προϋποθέσεις ασφαλείας ε, όσον αφορά στην κατάσταση στη Συρία. Και στο ερώτημα για το ρόλο του Κατάρ και τη στήριξη του Κατάρ στην Αλ-Νούσρα, δυστυχώς αυτός που είπε ότι το Κατάρ στηρίζει την Αλ-Νούσρα έχει ψευδίσει εσφαλμένες πληροφορίες. Εμείς δεν στηρίξαμε ποτέ την Νούσρα, στηρίξαμε τη μετριοπαθή αντιπολίτευση και έχουμε και άλλους Ευρωπαίους εταίρους στο πλευρό μας. Η Σαουδική Αραβία, διάφοροι άλλοι περιφερειακοί εταίροι, Ευρωπαίοι εταίροι και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, είχαμε συναντηθεί σε, μια αίθουσα επιχειρησιακή όπου διοχετεύσαμε και τη στήριξή μας. Ορισμένα μέσα μαζικής επικοινωνίας που έχουν επηρεαστεί από αυτή την εκστρατεία προπαγάνδα σε βάρος της χώρας μου ε, ξεκίνησαν αυτή την κρίση και διέδωσαν αυτές τις πληροφορίες. Ελπίζουμε όλοι να το ερευνήσουν περισσότερο το θέμα και να καταλάβουν ότι το, το Κατάρ ποτέ δεν ανέχθηκε και δεν στήριξε ακραίες εξτρεμιστικές ομάδες. Ποτέ δεν στηρίξαμε ανθρώπους που επιβάλλουν την υποταγή στην Αλκάιντα και στο Νταέσ. Αυτοί μάλιστα θεωρούν τις μουσουλμανικές χώρες ως προδότες. Και για εμάς αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη απειλή. Ξέρουμε ότι τελικά αυτές οι ριζοσπαστικές και ακραίες ομάδες θα στραφούν εναντίον μας ως μουσουλμανικές χώρες. Το αναγνωρίζουμε και γι' αυτό εργαζόμαστε στρατηγικά για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια που θα, που θα διοχητεύονται προς τις τρομοκρατικές δράσεις. Όταν τελικά δίνω ευκαιρίες σε παιδιά να ξαναμπούν στο σχολείο και να έχουν εκπαίδευση και να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα ίδια και για την ευρύτερη περιοχή. Αυτό κάνω. Αντικαθιστώ το όπλο με το μολύβι. Και αυτή είναι και η καλύτερη γιατριά. Τώρα, ως προς το Ιράν, σίγουρα υπάρχουν διαφορές. Όμως διαφορές οι οποίες δεν είναι ε, καθοριστικές. Θα λυθούν και λύνονται μόνο μέσα από ένα διάλογο άμεσο, απευθείας δεν πρέπει να έχουμε συνεχώς ε, ε, πλήρη εξουσίους και να κάνουμε διάλογο μέσω αντιπροσώπων και μέσω άλλων, γιατί το τίμημα το πληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Στην Ιεμένη βλέπουμε τα δυνατά αποτελέσματα. Ήμασταν μέρος του συνασπισμού της Συμμαχίας το 2015, ο οποίος είχε ως στόχο να επιφέρει πολιτική λύση σε αυτή τη διένεξη και να κάνει τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Συνεργασίας του, του Κόλπου πραγματικά να συνεργαστούν. Και τώρα έχουμε βασανιστήρια, έχουμε διαφορετική ατζέντα από κάθε ένα από τα μέλη τους της συμμαχίας. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος και δεν υπάρχει πολιτική στήριξη. Το Κατάρ δεν θα στηρίξει ποτέ τη θέση του Ιράν ή οποιοδήποτε άλλο για τη θέση για τον πόλεμο στην Ιεμένη. Εμείς στηρίζουμε την άποψη σύμφωνα με την οποία ο λαός της ε, Ιεμένης πρέπει να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων εκεί να βρουν μια λύση να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι. Είναι μια θαυμάσια χώρα η οποία όμως βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής η Ιεμένη. Ε, δέκα εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από ασυτεία και υποψήφια θύματα είναι άνω των 8 εκατομμυρίων στα τέλη αυτής της χρονιάς. 20 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από τις καταστραταγήσεις και παραβάσεις του διεθνούς δικαίου. Και η διεθνής κοινότητα το μόνο που κάνει είναι να καταδεκάζει στα λόγια. Πρέπει να αναλυφθούν ε, δράσεις. Να επιστρέψουν όλοι στο δρόμο της λογικής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήρθατε. Ευχαριστούμε για την ανταλλαγή απόψεων. Πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή για τα μέλη της Επιτροπής. Γνωρίζετε ότι το Κατάρ έχει πολλούς φίλους σε αυτή την Επιτροπή. Εμείς όμως παραμένουμε ουδέτεροι στην κρίση του κόλπου. Και αυτό βεβαίω που θέλουμε είναι να υπάρχει ενότητα στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, και βεβαίως θα θέλαμε να προσκαλέσουμε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Υποπιτροπή ή άλλες επιτροπές να έρθετε σε εμά να δείτε ποιο είναι αυτό το οποίο μιλάμε και παρουσιάζουμε το όραμά μας, να τα δείτε επιτόπου, στην πραγματικότητα και όχι απλά θεωρητικά. Ευχαριστούμε πολύ. <laughs> Thank Ladies Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε 15 λεπτά καθυστέρηση και ε, θα ήθελα τώρα τους ε, φίλους του Κατάρ, οι δυνατόν να αποχωρήσουν ήσυχα από την αίθουσα και να περάσουμε second try. Λοιπόν, ε, περνάμε στο επόμενο θέμα, το 18α που συμφωνήσαμε να το συζητήσουμε χθε. Θα μιλήσουμε για τη Μολδαβία. Να πω λίγα λόγια στην αρχή για να μπορούμε κάπως να δομήσουμε τα επόμενα 30 λεπτά. Δύο θέματα έχουμε να εξετάσουμε. Πρώτον, τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα, κυρίως στο Κισινάι, στην ε, πρωτεύουσα. Αυτό μας επισημάνθηκε χθε. Και επίση ε, θα μιλήσουμε και για μια κοινοβουλευτική ερώτηση που εκκρεμεί. Την Τρίτη το βράδυ θα γνωρίζετε ότι το δικαστήριο της πρωτεύουσα αποφάσισε να μην επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα ε, των εκλογών της 1 η Ιουνίου και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Οστέβιτσους για να μας ενημερώσει καλύτερα. Και πριν δώσω το λόγο στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάσουν, θα ήθελα να αναφερθώ και στο δεύτερο θέμα, το οποίο ανέφερα προηγουμένως για να τα συζητήσουν και τα δύο. Στις 21 Μαρτίου ο κύριος Σόλτς από την UNGL υπέβαλε μια κοινωνική ερώτηση στην Επιτροπή που αφορά στην ε, διερεύνηση οικονομικής απάτης στη Μολδαβία. Βασικά θα έπρεπε να απαντηθεί σε έξι εβδομάδες ε, αυτό το θέμα και μετά να τεθεί στη υπόψη μας. Έχουμε πέρασει τώρα περίπου τρεις μήνες και με βάση το 135 πράγματι το θέμα μπορούμε πλέον να το συζητήσουμε εμείς. Θα μιλήσουμε πρώτα για την Κίσινα, μετά για την ερώτηση του κυρίου Σόλτς και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάια Χάρτινγκ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι διευθυντής για την ε, Ευρώπη και την Ασία και η κυρία Ζιπάλα, η οποία είναι από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ε, βρήκατε χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας. Αν λοιπόν ισχύει αυτό και οι δύο δεσμευόμαστε στο να ε, εφαρμόσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης. Δηλαδή, εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθούμε και στηρίζουμε τη δημοκρατία της Μολδαβίας σε κάθε τη βήμα. Και από την άλλη πλευρά, εκείνοι δεσμεύονται στο να ε, καλύπτουν όλα τα οικονομικά και άλλα κριτήρια που είναι απαραίτητα για να ισχύει ένα συγκεκριμένο επίπεδο διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο δήμαρχος του Κισινάου, ο κύριος Κυρτουάκα, απομακρύνθηκε από το αξίωμά του, διότι κατηγορήθηκε για οικονομικές ατασταλίες και ανακοινώθηκαν, προκηρύχθηκαν νέες εκλογές. 20 Μαΐου, πρώτος γύρος, 1η Ιουνίου, δεύτερος γύρος των εκλογών έλαβαν χώρα στο Κισινάου. Προς μεγάλη μας λοιπόν έκπληξη, στις 19 Ιουνίου το δικαστήριο το τοπικό, το αστικό του Κισινάου ανέφερε ότι δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των ε, εκλογών και ε, μάλιστα είχε αναβάλει το θέμα για δύο φορές. Ως εκ τούτου, οι εκλογές που έλαβαν χώρα για τον νέο δήμαρχο του Κισινάου στις 19 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου δεν επικυρώνονται και μάλιστα ο Αντρέι Ναστάση, ο εκλεγμένος πλέον δήμαρχος, ο οποίος εκπροσωπεί την πλατφόρμα την φιλοευρωπαϊκή, αυτός δεν ε, επιβεβαιώθηκε στο αξίωμά του. Να επενθυμίσω όμως ότι ε, ο Αναστάση συγκέντρωσε το 52% των ψήφων στις 3 ε, Ιουνίου και κατανίκησε ε, τον υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με βάση την κοινή δήλωση που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Επιτροπή συγκεκριμένα στις 13 Ιουνίου του περασμένου έτους, με βάση λοιπόν αυτή τη δήλωση και παρατέτω. Λαμβάνω υπόψη των πρωτοβουλειών που έχουν αληθεί για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπής ανέφερε ότι μία προϋπόθεση, ένα προαπαιτούμενο για να χορηγηθεί οικονομική βοήθεια είναι η χώρα να έχει δημοκρατικό μηχανισμό, ε, πολυκομματική μορφή διακυβέρνηση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η ε, Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης θα ελέγξει την υλοποίηση αυτών των προαπαιτούμενων ε, για να μπορεί να εκταμιευτεί οικονομική βοήθεια και συνεχίζει πιο κάτω η ανακοίνωση. Αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι με αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία δεν αμφισβητώ, αλλά θέλω να εξηγήσω λιγάκι την περιραίουσα ατμόσφαιρα όπου ελήφθη αυτή η απόφαση, πολλοί κατέβηκαν στους δρόμους της Κισινάου εχθές, δεν ξέρω βέβαια πόσο ε, θα συνεχίσουν να διαδηλώνουν, αλλά θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση για να έχουμε αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ότι πράγματι γίνονται σεβαστά τα πολιτικά κριτήρια και εφαρμόζονται πλήρως την ε, δημοκρατία της Μολδαβίας Αυτά για να έχουμε μια καλή έκθεση σχετικά με τη δημοκρατία της ε, Μολδαβίας. Είπαμε αυτό να γίνει μέχρι τις τερνές ε, διακοπές. Το θέμα θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια η δημοκρατία της ε, Μολδαβίας ε, πρέπει να καλύπτει αυτά τα πολιτικά κριτήρια για να δεχτεί ε, χρηματοδοτική βοήθεια εν ευθέτω χρόνο. Και θέλω να επισημάνω ότι στις 26 Φεβρουαρίου του 2018 το Συμβούλιο αυτό για άλλη μια φορά κατέληξε σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Απλά να σας υπενθυμίσω παράγραφος 19 και παράγραφος 24. Εκεί αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι είναι πρόθυμη να στηρίξει τη δημοκρατία της Μολδαβίας με βάση συγκεκριμένη και ικανοποιητική πρόοδο σε όλους τους τομείς των μεταρρυθμίσεων και με βάση αυστηρά κριτήρια και προαπαιτούμενα. Κύριε Πρόεδρε, με όλα αυτά κατά νου θα πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο για να αναλύσουμε ε, την ε, ε, απόφαση του δικαστηρίου, το αιτιολογικό της απόφασης. Χρειαζόμαστε χρόνο βέβαια γι' αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να πολιτικοποιήσουμε το θέμα γιατί μιλάμε για το κράτος δικαίου και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Θέλω όμως να ακούσω κάποια σχόλια από την αρμόδια γενική διεύθυνση για να μας πει πώς ακριβώς ε, το θέμα αυτό της απόφασης του δικαστηρίου ε, συμβαδίζει με την τήρηση των προαπαιτούμενων. Και πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, ε, το οποίο θα ζητήσουμε σήμερα. Το λόγο έχει ο κύριος Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ. Όπως μας είπατε και προηγουμένως, ζήτησα γραπτή απάντηση όσον αφορά την ενδεχόμενη οικονομική απάτη στην οδηγία, στην Δημοκρατία της ε, Μολδαβίας. Ε, θα επαναλάβω λοιπόν ε, τα γεγονότα. Στο τέλος του 2014 ένα δις δολάρια αφαιρέθηκαν, μετακινήθηκαν από τις τράπεζες της Μολδαβίας. Όμως τα χρήματα αυτά ε, φαίνεται ότι εκλάπησαν και ότι δεν ε, επέστρεψαν ποτέ στην ε, τράπεζα. Έγιναν εσωτερικές έρευνες τμήματα των οποίων έχουν δημοσιευθεί, δεν έχει δημοσιευθεί όμως το σύνολο, αλλά το 2017 φάνηκε ότι τουλάχιστον 50% των ε, χρημάτων έχουν δοθεί ε, σε χώρες ε, που δεν είχαν δικαίωμα. Αναρωτιόμαστε λοιπόν σε ποιο βαθμό υπάρχει συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου και στις υπόλοιπες χώρες και ε, θέλουμε να ξέρουμε εάν ε, το μήμα των χρημάτων αυτών ε, αφορά και χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπλέκεται και η Κρόλ και θα θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται. Επίσης, ε, πιστεύει η Κομισιόν ότι ε, υπάρχει κάποια νομική βάση έτσι ώστε ε, να μπορέσει μετά από αυτή την κλοπή και λόγω των νομικών προϋποθέσεων να μπλοκάρει κάποια χρήματα και εν πάση περιπτώσει ποια δράση έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και απέναντι στην Ουκρανία, το Χονγκ Κόνγκ και την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έτσι ώστε να βοηθήσουν ε, στην επίλυση της ε, κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα πλέον έχει μια πιο σαφή εικόνα από τους δικηγόρους στην Μολδαβία ότι οι αρχές επιβολής του νόμου δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους έτσι ώστε να ε, ε, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης η Όλαφ μελε... ερευνά το θέμα ή κάποιες άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερευνούν το θέμα των χρημάτων αυτών που αφαιρέθηκαν από την τράπεζα, από τις τράπεζες. και ε, ε, ε, υποβάλλει προϋποθέσεις σχετικές με την υπόθεση αυτή στην Δημοκρατία της Μολδαβίας. Ευχαριστούμε πολύ, Χελμούτ. Θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Μάια Χάτι. Καλωσορίσατε και ευχαριστούμε που ενώ σας ειδοποιήσαμε τελευταία στιγμή αποδεχτήκατε την, το αίτημά μας και είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι θα προσπαθήσω να απαντήσω στο γενικό ερώτημα για τις ε, εξελίξεις όσον αφορά την κατάσταση και μετά θα απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Σόλτ, αλλά αν και νομίζω ότι ίσω ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν θα θέλει να απαντήσει για το θέμα αυτό. Να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερική δράση παρακολουθούν από κοντά τι τελευταίε εξελίξει στην ε, δημοκρατία τη ε, Μολδαβία. Ε, η απόφαση του δικαστηρίου του Κισινάου να μην επικυρώσει το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών και την εκλογή του Δημάρχου του Κισινάου Προφανώ. Ε, μας προκαλεί ε, μεγάλο προβληματισμό και συζητήθηκε το θέμα, ε, να σας πω, και με την υπατή εκπρόσωπο χθες το βράδυ. Ο κύριος Νασταζέ, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, εξελέγει με πλειοψηφία που υπερβαίνει το 52% και αναγνωρίστηκε ως δήμαρχος και από τα, τους ξένους παρατηρητές, αλλά και από τον ιτημένο αντίπαλό του. Ε, πρέπει η δημοκρατία του, της ε, Μολδαβίας να σεβαστεί και τις, ε, τους διεθνείς όρους δικαίου αλλά και τους όρους της διμερούς συμφωνίας και οπωσδήποτε θα πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα με τρόπο σωστό, διαφανή και με σεβασμό της έκφρασης της βούλησης έτσι όπως αυτή εκφράστηκε μέσω των εκλογών των πολιτών της ε, Μολδαβίας να ε, υπενθυμίσω ότι οι ελευθερίες του ε, ε, συνεδριάζει και η ελευθερία συνέλευσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προσπαθούν να αναλύσουν την κατάσταση. Βεβαίως εμείς συνδυάζουμε και συντονιζόμαστε και με άλλους διεθνείς οργανισμούς και παρατηρητές. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ε, το, ε, ε, το θέμα της Μολδαβίας μας απασχόλησε πέρσι, οπότε και μεταρρυθμίστηκε το εκλογικό σύστημα. Ε, στο, στην κοινή δήλωση του Συμβουλίου της ε, Κομισιόν ε, που έχει προσαρτηθεί σε την απόφαση για μακροοικονομική αρρωγή αναφέρονται τα στοιχεία αυτά. Ε, και ε, είναι σαφές ε, ότι δεν μας ενδιαφέρει μονάχα η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση και σεβασμός των συμφωνηθέντων αλλά και ένα σωστό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό σύστημα το οποίο, το, οποίο ενστερνίζεται τα δημοκρατικά ιδεώδη και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τα τεκτενόμενα στη χώρα υπάρχει προβληματισμός και πρέπει πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά το θέμα και το κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί ε, και η μακροοικονομική αρρωγή. Η κατάσταση στην ε, ε, Μολδαβία έχει αλλάξει από πέρσι τον, το Συμβούλιο του Φεβρουαρίου του 2018 αναφέρθηκε στο θέμα της ε, Μολδαβίας. Έγιναν κάποιες, ε, τροποποιη, κάποιες μεταρρυθμίσεις, αλλά βεβαίως ε, όχι αυτές ε, που θα θέλαμε και στο βαθμό που θα θέλαμε. Όσον αφορά τώρα το θέμα της, ε, των ερευνών όσον αφορά την τραπεζική απάτη. Πρέπει να σας πω ότι για το θέμα αυτό ο προβληματισμός μας είναι πάρα πολύ μεγάλος ε, και σχετίζεται και με τον σεβασμό του κράτους ε, δικαίου στην δημοκρατία της Μολδαβίας. Για μία ακόμα φορά οι ευρωπαϊκές αρχές ζήτησαν επισταμένως από τις αρχές της Μολδαβίας να ερευνήσουν το θέμα με τρόπο ακέραιο και αντικειμενικό και αδέκα Ωστόσο, πιστεύουμε ε, ότι όντως ε, έχει ε, πάρει κάποια μέτρα η κυβέρνηση της Μολδαβίας αλλά παρόλα αυτά, και για να το πω πολύ προσεκτικά, δεν πιστεύουμε ότι τα μέτρα αυτά είναι αρκετά έτσι ώστε να αποτρέψουν ε, μια μελλοντική παρόμοια κατάσταση και δεν είναι σίγουρα ε, ικανά έτσι ώστε να εξηγιάνουν το τραπεζικό σύστημα. Ε, να σας πω ότι ο κύριος Νάσταζε είχε παίξει σημαντικό ρόλο στις διαμαρτυρίες που είχαν οργανωθεί με λόγω ακριβώς αυτής της τραπεζικής απάντησης ήταν τότε ηγέτης και της αντιπολίτευσης ε, στις κινητοποιήσεις αυτές ε, και ε, ενδεχομένως υπάρχει κάποια διασύνδεση ανάμεσα στον τρόπο αντιμετώπισης της τραπεζικής απάτης αφενός και την πολιτική κατάσταση όσον αφορά αυτόν τον δημοκρατικά εκλεγμένο δήμαρχο του Κισινάου. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ κύριε Μάιε Χάρτιν. Έχετε κάτι να προσθέσετε? Τότε να δώσω το λόγο στη DG Home. Η κυρία Σύπαλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε από τη DG Home και τη μετανάστευση. Δύο λόγια καταρχάς για να πω πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσιλωμένη προς μια ε, απάντηση υψηλής ποιότητας επί του προκειμένου στο ερώτημα το γραπτό που της απευθύνθηκε και γι' αυτό ε, πρέπει να έχουμε εσωτερική συνεργασία και εσωτερικό συντονισμό θα έχουμε επίσημη γραπτή απάντηση σε αυτό το πολύ σημαντικό ερώτημα ε, λίαν συντόμως, μόλις ολοκληρώσουμε τις ε, εσωτερικές μας διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το ζήτημα της μαζικής απάτης και των συνεπειών τους. Ο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ήδη ανέφερε το σχετικό σημείο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου του 2018. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι οι συνέπειες αυτής της απάτης γίνονται αντικείμενο αναφοράς στην αναθεωρημένη ατζέντα συνεργασίας για την ε, τριετία, αναθεωρημένη που υιοθετήθηκε τον Αύγουστο της περασμένης χρονιάς. Γίνεται ειδική μνήμα στην τραπεζική απάτη και στην ανάκτηση στοιχείων ενεργητικού. Ζήτα, ερωτάτε δύο, κάνετε δύο ερωτήσεις αξιότιμα μέλη. Πρώτον, ποια εργαλεία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει το θέμα της ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων και δεύτερον, ποια είναι η εμπλοκή και η συμμετοχή των ευρωπαϊκών φορέων και οργάνων. Έχουμε την οδηγία για την κατάσχεση του 2014 και με αυτή την οδηγία όλα τα κράτη-μέλη έχουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο ενσωματώνοντας την οδηγία στην εθνική τους ένωμη τάξη για να δεσμεύσουν και να κατάσχουν ε, τις προσόδους ε, που προέρχονται από το έγκλημα. Εάν λοιπόν υπάρχουν στοιχεία ενεργητικού, περισσοιακά στοιχεία που υπάρχουν στα κράτη-μέλη λόγω αυτής της τραπεζικής απάτης και αν αναγνωριστούν και εφόσον αναγνωριστούν ως τέτοια, τότε οι δικαστικές αρχές των κρατών μελών με βάση την εθνική νομοθεσία που έχει ενσωματώσει την οδηγία του 2014 για δίμευση και κατάσχεση έχουν τα κατάλληλα νομικά εργαλεία να αναλάβουν την κατάλληλη δράση. Αναφέρω το δίκτυο των γραφείων ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωση. όπου οι ε, κρατικές αρχές έχουν τη δυνατότητα μέσα από αυτό το δίκτυο να ανταλλάξουν πληροφορίες και να εντοπίσουν και να ανοιχνεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία ή τα στοιχεία ενεργητικού που πρέπει να δεσμευθούν ή να δημευθούν ή να κατασχεθούν. Αναλόγως ε, τι πρέπει να γίνει, ε, εμείς ενισχύουμε τη συνεργασία και την εθαρρύνουμε μεταξύ κρατών μελών έτσι ώστε να ανακτηθούν τελικά αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Βεβαίως όποιος υπονομεύει την έρευνα είναι υπόλογος και υπόκειται σε κυρώσεις βάσει εθνικής νομοθεσίας. Τώρα, αν εμπλέκεται η Europol και η Eurojust πρέπει να τις ρωτήσουμε και να σας ενημερώσουμε σχετικά κατά πόσο συμβάλλουν σε αυτές τις έρευνες και αυτά θα τα περιλάβουμε στη γραπτή μας απάντηση στο ερώτημα που μας έχετε απευθύνει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ για αυτά τα στοιχεία από το εκτελεστικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Πόσο χρόνο έχουμε? Δέκα λεπτά. Ο κύριος Πρέντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι σήμερα είμαστε σε θέση να συζητούμε για την ε, δημοκρατία της Μολδαβίας. Ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης μπορώ να σας μιλήσω ξεκάθαρα και να σας πω πώς βλέπω την κατάσταση των Μολδαβών πολιτών. Πώς αντιμετωπίζουν το θέμα επιτόπου. Όλοι ξέρουν ότι τη Μολδαβία την κυβερνάει ένας παρανοϊκός ολιγάρχης. Από τη μία έχουμε ένα δημοκράτη και έναν, απ' την άλλη ένα σοσιαλιστή. Ε, ε, το συγγνώμη, ένα, αυτοί οι δύο, ο Δημοκράτης και ο Σοσιαλιστής, έχουν μπλοκάρει την οικονομική βοήθεια. Έχουμε το Δημοκρατικό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα και τελικά το αποτέλεσμα ήταν τελείως διαφορετικό. Μπλόκαραν της έρευνας για αυτή την τεράστια τραπεζική απάτη. Αυτοί οι δύο ηγέτες των δύο ε, πολιτικών κομμάτων, του Δημοκρατικού και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, προσπαθούν να ακυρώσουν και τα αποτελέσματα των δημοκρατικών εκλογών του Κίζινάου. Όλοι το ξέρουν και όλοι το βλέπουν. Στις Βρυξέλλες τώρα εδώ γίνονται απόπειρες να αποκριβεί αυτό το γεγονός. Κάποιοι παρουσιάζουν τον Ρεντνούκ ως ήρωα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως έχει απόλυτη επικυριαρχία στη Μολδαβία, Μολδαβία και αυτή την έχει χάρη στη στήριξη των κομμουνιστών βουλευτών. Πιστεύω ότι είναι πολιτικό το πρόβλημα και πρέπει να ακούσουμε τον λαό της Μολδαβίας, τους Μολδαβούς πολίτες και όχι αυτούς που διαδίδουν ε, προπαγανδιστικά εσφαλμένες ειδήσει. Η κατάσταση λοιπόν έχει ως εξής έχουμε επέκταση της πολιτικής ενός κόμματος, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της ε, ε, Ρουμανίας, που είναι άμεσα υπεύθυνο για την έλευση αυτής της κρίσης στη δημοκρατία της Μολδαβίας. Προσπάθησε να πείσει τα κρατη και τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Σοσιαλδημοκρατικό αυτό κόμμα, ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ δημοκράτη και σοσιαλιστή είναι προϊόν ευγενούς άμυλας. Όμως αυτό είναι ψευδές, είναι εσφαλμένο. Πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετηθούν ξεκάθαρα μέτρα, σοβαρά μέτρα, γιατί λέγονται πάρα πολλά ψέματα αυτή τη στιγμή στη Μολδαβία. Να ξεκαθαριστεί το θέμα της ε, ε, χρηματοοικονομικής βοήθειας, να μπορέσουμε να έχουμε μια δημοκρατία που να λειτουργεί. Δηλαδή, να σεβόμαστε τη βούληση των πολιτών και να παρετηθούμε από τις ψευδεστήσεις μας για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται αυτή η χώρα, για να μπορέσει ο λαός της Μολδαβίας να έχει μια ευκαιρία για το μέλλον. Ευχαριστώ τον κύριο ε, Πρέντα, ο κύριος Μποστινάρου για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σχολιάσω τους ισχυρισμούς του κυρίου Πρέντα, διότι είναι αβάσιμοι οι ισχυρισμοί αυτοί και σας καλώ να δείτε τα γεγονότα και θα αναφερθώ αποκλειστικά και μόνο στα γεγονότα. Γιατί έστω και αν ορισμένοι από τους ισχυρισμούς του κυρίου Πρέντα ε, ε, είχαν κάποια βάση, θα ήμουν ο πρώτος που θα ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εσάς να αναθεωρήσετε τις σχέσεις σας με τη Μολδαβία. Ποια είναι λοιπόν τα γεγονότα. Είναι μια πολύ ανησυχητική απόφαση και δεν είναι δίκαιο να σχολιάζει κανείς τις αποφάσεις του δικαστή. Ωστόσο, πολιτικά μας σημαίνει το καμπανάκι του συνεγερμού και αναφέρομαι στην πολιτική δήλωση του κυρίου Ναστάση, μια πολιτική απόφαση που λαμβάνει δικαστής, ο οποίος περιφρόνησε όλους εμάς σήμερα και περιφρόνησε και την ε, βούληση της κοινή γνώμης και ε, προσυπογράφω πλήρως αυτή τη δήλωση και την στηρίζω απολύτω. Όμως, από την απόφαση αυτή μέχρι τον ισχυρισμό ότι αξιοποιήθηκε δικαστική εξουσία ως πολιτικό όργανο από ορισμένου πολιτικούς ή από την κυβέρνηση στο Κιζινάου, η απόσταση είναι μεγάλη. Δεν θέλουμε να διαδίδονται ισχυρισμοί χωρίς να συνοδεύονται από στοιχεία. Ποια είναι τα γεγονότα για να καταλάβετε κι εσείς περί τίνος πρόκειται. Η απόφαση εξυπηρετεί το Δημοκρατικό Κόμμα. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν, την δεν το εξυπηρετεί, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δεν έχει άμεσο υποψήφιο για το ΚΙΖΙΝΑΟ... Και στο δεύτερο γύρο ρητός εξέφρασε το Δημοκρατικό Κόμμα τη στήριξή του στον κύριο Ναστάσε. Και σας καλώ αυτό να το παληθεύσετε και να το εξακριβώσετε. Υπήρξε επίσημη συνάντηση μεταξύ της ηγεσία της κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Κόμματος με τους πρέσβεις στο Κιζινάο, παρουσία του Αμερικανού πρέσβη, και εκεί του ζητήθηκε με κατά κάποιο τρόπο να παίξουν το ρόλο του πληροφορία δόθηκε αγγελιοφόρου προς τον κύριο Ναστάσε και να ρωτήσουν τον κύριο Ναστάσε ως αγγελιοφόροι υπό ποιε προϋποθέσεις και ποια είδους πολιτική στηρίξη θα ήθελε για το δεύτερο γύρο για να μπορέσουν να την εγγυηθούν αυτή την πολιτική στήριξη και το μήνυμα αυτό διαβιβάστηκε στον κύριο Ναστάσε και μάλιστα στο δεύτερο γύρο και στις εκλογές ε, έγινε αυτό που συνέφερε τον κύριο Ναστάσε έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό μου το Κίζι Νάου έχει ένα δήμαρχο υπέρ της Ευρώπης και όχι ένα δήμαρχο σοσιαλιστή. Και μάλιστα αυτό συνέβη όχι χωρίς σημαντική συνεισφορά από τη δική μας πλευρά. Ήταν μήνυμα στο κινητό από κάποιον από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από το Κοινοβούλιο να επαληθεύσουν, να εξακριβώσουν με όλους τους δυνατούς τρόπους ποια είναι τα προβλήματα, πώς μπορούμε να προσφύγουμε και να αποκατασταθεί η κατάσταση για να μην υπάρξει ξέσπασμα πολιτικής κρίσης και να επικρατήσει ηρεμία στο πολιτικό σκηνικό για να μπορέσουν να διεξαχθούν ομαλά κοινοβουλευτικές εκλογές. Με αυτή την κατάσταση δύο είναι μόνο οι νικητές, ο κύριος Ντοντών και η Ρωσία. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ η Ρεμπέκα Χάρμς, τελευταία ομιλήτρια. Παρακαλώ. Έχω να υποβάλω άλλες δύο ερωτήσεις ε, και θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον αυτές οι τοπικές εκλογές, ε, κατά πόσον σε αυτές τις εκλογές υπήρχαν, ε, υπήρχε ομάδα παρακολούθηση των εκλογών. Και θα ήθελα να γνωρίζω και τη σύνθεση του εκλογικού συμβουλίου του Κισινάου. Γιατί αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν καταφύγει στο δικαστήριο. Και πέρα από αυτά τα δύο, Νομίζω ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι κατανοώ απόλυτα γιατί ο κυρίος Οστρεβίτσιους συνδέει όλα αυτά που συζητάμε για τη Μολδαβία με τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στη χώρα. Από την άλλη βέβαια θα ήθελα να ενσκύψουμε στην ουσία του προβλήματος γιατί στη Μολδαβία υπάρχουν δυσλειτουργίες του συστήματος και σε τελική ανάλυση ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα που θα είναι και ακριβό οι απλοί πολίτες της ε, Μολδαβίας. Γιατί δεν θα υπάρχει καμία πρόοδος ε, σε αυτή την απάτη του αιώνα στη Μολδαβία και πλέον όλα τα προβλήματα προκύπτουν μετά ε, την εκλογή ενός δημάρχου ο οποίος είναι φιλοευρωπαίος, ο οποίος είναι κατά της διαφθοράς και ο οποίος είναι σαφώς κατά των ολιγαρχών της Μολδαβίας. Δεν ξέρω τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε και εμείς ε, να προσφύγουμε κατά της απόφασης του δικαστηρίου, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία προσφυγή και όλοι στη Μολδαβία οφείλουν να κατανοήσουν ότι εμείς εδώ στις Βρυξέλλες δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτά που διαδραματίστηκαν εκεί, όχι γιατί απλά η Μολδαβία βαδίζει στο δρόμο των εθνικών εκλογών μέχρι το τέλος του έτους και όλα τα προβλήματα που βλέπουμε τώρα ε, ενδέχεται να επανέλθουν και στις εθνικές εκλογές. Και αρκετές συζητήσεις είχαμε με τους συναδέλφους μας από τη Μολδαβία για τα προβλήματα που υπάρχουν στην ε, μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Υπάρχει και το θέμα της δίκης αντιμετώπισης στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης με βάση αυτή την ερώτηση που συζητάμε. Όλα αυτά συνδέονται με όσα διαδραματίστηκαν πριν από λίγες ημέρες στο Κισνό, αλλά εμείς όλα αυτά τα συζητάμε εδώ και πολύ καιρό και ειλικρινά δεν έχουμε δει καμία απολύτως βελτίωση. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χάρμς, ήταν σαφέστατη στην παρέμβασή της. Ήδη έχουμε καθυστερήσει ένα τέταρτο. Λίγα λεπτά θα έχετε για να απαντήσετε στους ερωτώντες, τους τρεις και Νομίζω μου είπαν ότι έχουμε και τον κύριο Λένατς ε, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση οικονομικής βοηθείας. Αν θέλετε και εσείς ίσως μπορείτε να παρέμβετε. Λοιπόν, παρακαλώ πρώτα εσείς ή μάλλον ο άλλος κύριος από τη Γενική Διεύθυνση θα λάβει πρώτος το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας, δηλαδή την εκταμίευση των δόσεων, υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που είναι σημαντικά. Πρώτον, θετική αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής και των προποθέσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Δεύτερον, θα πρέπει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τρίτον, τα πολιτικά προαπαιτούμενα που αναφέραμε σήμερα το πρωί θα πρέπει και αυτά να πληρούνται. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε μαζί ε, με τις αρμόδιες υπηρεσίες το τι γίνεται με αυτά τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των δόσεων. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ορισμένα εξ αυτών ε, συνδέονται στενά με αυτά τα θέματα που συζητήθηκαν σήμερα εδώ. Τρία έχουν σχέση με την καταπολέμηση διαφθοράς και το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, αυτά τα προπετούμενα έχουν στόχο να προσφέρουν λύσεις στη Μολδαβία, διαρθρωτικής φύσεως, και έχουν στόχο τη σύσταση θεσμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος δηλαδή. Το θέμα είναι αυτοί οι θεσμοί να μπορούν να λειτουργήσουν. Μιλάμε για το θεσμό, το γραφείο ε, της ε, καταπολέμησης διαφθοράς και το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος που συστήθηκε πρόσφατα και επίσης και αυτό άλλαξε κάπως ε, αρμοδιότητες και λειτουργία. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με την πρόσληψη επιθεωρητών ελέγχου και έχουμε και έναν τρίτο νόμο για την ανάκτηση κεφαλαίων, ένα νόμο ο οποίος έχει ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία και την παροχή επαρκών ε, οικονομικών πόρων. Θα ξέρετε ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια νέα πολιτική ανάκτησης κεφαλαίων. Εδώ ο ρόλος του νέου φορέα είναι καθοριστική σημασία. Άρα δηλαδή αυτά που προβλέπουμε εμείς στο μνημόνιο ήταν θετικά, επικοδομητικά. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι όσον αφορά την τρίτη δόση προβλέπεται μια δράση που έχει άμεση σχέση με την τραπεζική απάτη και εκεί αναφέρεται ότι για να επανέλθουν στην τράπεζα ε, τα κεφάλαια τα οποία ε, διοχετεύτηκαν εκτός της χώρας ε, ε, μέσω απάτης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η στρατηγική που έχει καθοριστεί για αυτή την υπόθεση. Να πω λοιπόν ότι εμείς ε, έχουμε τονίσει ότι για να εκταμιευτεί η δόση αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εδώ θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου. Ε, παρακαλώ, έχετε και εσείς τη δυνατότητα να παρέμβετε. Μισό λεπτό. Ερώτηση θέλετε να υποβάλλετε. Ο κύριος Σόλτς μπορεί να σχολιάσει, είναι εντάξει για σας, παρακαλώ. Αλλά αν έχετε την καλοσύνη να είστε σύντομος γιατί δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, Άκουσα τις απαντήσεις ε, και ελπίζω η διαβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα δώσει σε μένα συγκεκριμένες απαντήσεις ε, για τις ερωτήσεις που έχω θέσει. Αυτό ελπίζω να γίνει όχι μετά από άλλους τρεις μήνες, αλλά ως το δυνατόν ταχύτερα. Και κατά δεύτερον, το θέμα το έχουμε ήδη συζητήσει. Έχουμε μιλήσει την τελευταία φορά για την παροχή οικονομικής βοήθειας στη Μολδαβία. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει γίνει. Άρα δηλαδή πρέπει να αλλάξει αυτή η στάση και θέλω να πιστεύω ότι ε, θα μας προσφέρετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούμε ε, αργότερα ενδεχομένω να επανέλθουμε στο θέμα. Πρόεδρος, εγώ έχω το πρόβλημα να χειρίζομαι σωστά αυτέ τι συζητήσει. Έχουμε ήδη καθυστερήσει 20 λεπτά. Ο κύριο Χάρτινγκ ε, θα ολοκληρώσει την παραμεστή και μετά δεν θα δεχτώ καμία άλλη παρέμβαση επ' αυτού. Ε, πρώτα απ' όλα, Επιτρέψτε μου να πω ότι όσον αφορά την οικονομική βοήθεια, εκπρόσωπος του, της Διεύθυνης ΕΚΦΗΝ αναφέρθηκε και στις οικονομικές ε, και πολιτικές ε, δεσμεύσεις. Να πω ότι όσον αφορά τα πολιτικά προαπαιτούμενα, λαμβανωμένο υπόψη των τελευταίων εξελίξεων, προφανώς και θα πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, τις εξελίξεις για να μπορούμε να καταλήξουμε σε μια τελική άποψη που θα επηρεάσει την οριστική απόφαση. Ε, υπάρχει αυτή η διαδικασία κατάθεσης προσφυγών και αυτή είναι καθοριστική σημασία. Να σας πω όμως ότι δεν είναι φυσικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για άλλους να ε, κρίνουν δικαστικές αποφάσεις. Από την άλλη πρέπει να πούμε ότι πράγματι η Μολδαβία έχει μια πολύ ατυχή παράδοση, δηλαδή την πολιτικοποίηση της δικαιοσύνη. και γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα πολύ προσεκτικά. Όπως είπα στην παρέμβασή μου, η, θέληση, η βούληση των ε, ψηφοφόρων του εκλογικού σώματος ε, είναι θέσφατο, δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτήν. Για τις άλλες παρατηρήσεις να σας πω ότι όσον αφορά την παρακολούθηση των εκλογών, τοπική ήταν, εξ όσων γνωρίζω, ε, θα πρέπει να επανέλθω όμω για το θέμα τη παρακολούθηση των εκλογών, να απαντήσω πώ ακριβώ είχε οργανωθεί η παρακολούθηση των εκλογών. Και για τι επιπτώσει. να πω ότι η δική μα η αντιπροσωπεία προσπαθεί με κόπο να βρει τι ακριβώ γίνεται με τον εκλογικό νόμο και με την απόφαση της δικαιοσύνη. Ε, καταλήξαμε στο ότι αυτή τη στιγμή δήμαρχος είναι η κυρία Ράντου, η οποία είναι ανεξάρτητη. Αλλά εξ όσων γνωρίζουμε πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα και όσο δεν έχει εκλεγεί εκλεγεί νέος δήμαρχος θα παραμείνει στη θέση της δημάρχου. Ε, οι νέες εκλογές θα λάβουν χώρα ανάλογα και με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Έχουμε δει κάποια ανάλυση ότι θα πρέπει να καθυστερήσουν οι επόμενες εκλογές μέχρι την επόμενη χρονιά. Άρα δηλαδή η κυρία Ράντιο θα παραμείνει στο αξίωμα της Δημάρχου για άλλο ένα χρόνο και αυτά είχα να σας πω. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτα άλλο επί του θέματος. Συνάδελφοι, για να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα εγώ ε, θα δημοσιοποιήσω μία δήλωση από κοινού με την κυρία Χάνς που είναι η συμπρόεδρος της Euronest και τον εισηγητή τον κύριο Στέβιτσους για τις εξελίξεις στη Μολδαβία θα αναφερούμε ότι είμαστε υπέρ των δημοκρατικών αρχών, ε, να μην υπάρχει καμία πολιτική παρέμβαση στη δικαιοσύνη και ε, θα τοποθετηθούμε και στο θέμα των εκλογών. Μετά ο εισηγητής μας θα πρέπει να μας ενημερώσει για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης Μολδαβίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος κ. Ντοντών έρχεται στις Βρυξέλλες και ζήτησε να συναντηθεί όχι μόνο με μέλη της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, 28 Ιουνίου θα έχουμε μια σύντομη συνάντηση μαζί του και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να επαναφέρουμε και κάποιες απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα. Πολύ ωραία, σας εύχομαι μια θαυμάσια ημέρα. So, where are our guests? Eric, are coming upstairs? So. Λοιπόν, η επόμενη προσκεκλημένη μας είναι ο κύριος Κούνιχ και So, dear colleague. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε στο σημείο υπαριθμών 19, που είναι και το τελευταίο θέμα της ημερήσια διάταξης για σήμερα, ανταλλαγή απόψεων ε, για την αποτροπή κρίσεων, τη σταθεροποίηση και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά όλα γίνονται και με τη συνεργασία της ομάδας DEG. Θα ήθελα πολύ θερμά να ε, καλωσορίσω τον κύριο Κιόνιχ. Ε, σας καλωσορίζουμε θερμά, Γενικό Διευθυντή ε, για την αποτροπή κρίσεων, σταθεροποίηση οικοδόμηση ειρήνη και μετά από συγκρούσει και την παροχή Ανθρωπικής Βοήθειας Γερμανικό Μοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών και ο κύριο Στεφάνο Τόματ, Επικεφαλής του Τιμάτος Πρίσμα Αποτροπή Συγκρίσεων Κράτου Δικαίου Ήδη έχουμε καθυστερήσει και θέλω πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Θα δώσω το λόγο στο Γερμανό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Κιούνιχ. Βεβαίως ε, ε, υπάρχει κάποια ζωφερή ατμόσφαιρα. Η ε, όλη η κατάσταση για την πρόληψη των κρίσεων έχει ήδη ε, αναλυθεί από την γερμανική κυβέρνηση και το ερώτημα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διοργανική συνεργασία όπως και τη συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έτσι ώστε να μπορούμε να βασιστούμε στις βέλτιστες δυνατές πληροφορίες, στους καλύτερους εμπειρογνώμονες και κύριε Τόματι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία και μόνο φωνή με βάση το σχέδιο του 2009 ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα μεγάλο βαθμό ευελιξία στις ε, διαπραγματεύσεις και στο να ε, ανακαλύπτει νέες οδούς. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώ μπορεί να γίνει με την ευελιξία όταν πρόκειται για τη διαμεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Κιόνιχ, μετά στον κύριο Τόματ και ελπίζω να μείνει και λίγο χρόνο για ερωτήσει από συναντέλφου. Σα. παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Okay. Well, thank you very much, Mr. And... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση που μου αποστήλατε έτσι ώστε να συζητήσω μαζί σας αυτά που κατά την άποψή μας είναι πολύ σοβαρά θέματα. Ε, όπως είπε και ο πρόεδρος σας ε, μόλις, την προηγούμενη χρονιά ε, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε νέες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την αποτροπή κρίσεων και την ε, σταθεροποίηση και αυτό αποτελεί ένα στρατηγικό έγγραφο μεγάλη σημασία για τη γερμανική κυβέρνηση, επί του οποίου προσπαθούμε και δια του οποίου προσπαθούμε να βρούμε καλύτερες λύσεις όσον αφορά την αποτροπή αλλά και την επίλυση ε, κρίσεων και συγκρούσεων. Πρόκειται για ένα ε, έγγραφο το οποίο ε, και ένα μέσο το οποίο ε, ενδυναμώνει τα μέσα τα οποία ήδη έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Ε, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες της εθνικής κυβέρνησης σε περιπτώσεις αντίδρασης κρίσεων και σε κρίσεις και συγκρούσεις. Η διαχείριση κρίσης, η πρόληψη κρίσεων, η διαχείριση, η επίλυση κρίσεων. Ό,τι θέλετε ε, επιλέξτε πάντα, πάντα δεν μπορεί η διαδικασία αυτή να αφορά ένα μόνο μέσο, ένα μόνο εργαλείο. Ε, πρέπει οπωσδήποτε και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε είναι μια προσέγγιση η οποία πρέπει να αφορά όλα τα Υπουργεία ε, και το σύνολο της ε, κυβέρνησης, τουλάχιστον ε, αυτό πιστεύουμε εμείς στη Γερμανία. Δεύτερον, αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση κατά την οποία έχουμε όλο ένα αυξανόμενο αριθμό συγκρούσεων και όλο ένα και μικρότερο αριθμό επιλύσεων συγκρούσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε αναλάβει ε, μία σε βάθος αναθεώρηση των ε, γερμανικών ε, πολιτικών. Όταν ξεκίνησε τη δεύτερη του θητεία ο Υπουργός Στάιν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και εκεί βρίσκονται οι ρίζες αυτής, αυτού του εγγράφου που σας αναφέρω εδώ. Ε, θέλουμε ε, και στόχος μας ήταν η συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων ε, σε δομικό, διαθρωτικό τρόπο, αλλά και μέσω συνεργασίας όλων των μέσων και εργαλείων που έχουμε στην διάθεσή μας, έτσι ώστε όλοι να αντιμετωπίζουν μέσα από μια κοινή αντίληψη το θέμα της διαχείρισης και επίλυσης των συγκρούσεων. Ένα βασικό στοιχείο ε, κατά την άποψή μας ε, στην αντίδραση ε, όσον αφορά κρίσεις και συγκρούσεις και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο. Αυτό που προσπαθούμε δηλαδή ως Γερμανία να κάνουμε όταν αντιδρούμε σε κάποια κρίση είναι να πούμε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και μια πολιτική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί η ιδέα, το πλαίσιο ε, των όσων θα θέλαμε να ε, επιτύχουμε σε συγκεκριμένες συγκρούσεις και κρίσεις. Αυτό ξεκαθαρίζεται πρώτα και μετά προχωράμε στους τρόπους με τους οποίους η διαδικασία θα προχωρήσει και ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία ή οι διαδικασίες αυτές θα ολοκληρωθούν. Βέβαια αυτό το λέει κανείς ευκολότερα από ότι το κάνει γιατί ε, στην πράξη δεν είναι τόσο απλό. Ε, πρέπει βεβαίως ε, να μάθει κανείς να δουλεύει και σε διακυβερνητικό επίπεδο ή μάλλον ενδο κυβερνητικό επίπεδο. Πολλές συζητήσεις γίνονται γύρω από το τραπέζι μέχρι να αποφασιστεί μια κοινή στρατηγική μέχρι ότου ρυθμιστούν λεπτομέρειες κοινών επιχειρήσεων. λέω ότι ένας νόμος μόνος του ε, και από μόνος δεν μπορεί να λύσει μια κρίση ε, και κατ' επέκταση μια χώρα μόνη της δεν μπορεί να επιλύσει μια κρίση. Αυτό που βλέπουμε και μας ε, χαροποιεί ιδιαιτέρως ε, είναι ότι διαπιστώνουμε ότι σε πολλά επίπεδα οι διεθνείς εξελίξεις ε, ακριβώς υποβάλλουν τα ίδια ερωτήματα και επιζητούν παρόμοιες λύσεις ίσως από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και το σημαντικό είναι η οικοδόμηση συμμαχιών. Για παράδειγμα, από τότε που βρέθηκα στο κέντρο, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει τα ίδια ερωτήματα και ε, επιλέγει την ε, integrated approach, την ολοκληρωμένη προσέγγιση, που ακριβώς αυτή χρειάζεται. Έχουμε νέες υπηρεσίες, όπως ας πούμε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχουμε άλλωστε τον συνάδελφο, τον ε, Στεφάνο, που είναι ακριβώς εδώ δίπλα μου και που εκπροσωπεί την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ε, είναι σημαντικό να βλέπουμε τι μέσα, τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας, πώς μπορούμε ε, από κοινού να βάλουμε στην υπηρεσία της επίλυσης ή διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων αυτά τα εργαλεία. Επίσης, ε, ο Αντώνιο Γκουτιέρες, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ε, ε, καταβάλει μεγάλες προσπάθειες στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας και προσπαθεί να δημιουργήσει συνέργειες από την δική του την πλευρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό Τέλος, ε, όσον αφορά την διεθνή σκηνή, θα ήθελα να αναφερθώ στην Παγκόσμια Τράπεζα, ε, η οποία έχει διέλθει τα τελευταία χρόνια μέσω σημαντικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και έχει δημιουργήσει ε, μία μονάδα η οποία έχει τον τίτλο «Επίλυση βίας και συγκρούσεων». Υπάρχουν λοιπόν πολλά εργαλεία έτσι ώστε να ανταποκριθεί κανείς, να αντιδράσει ε, σε καταστάσεις ε, κρίσης ε, και είναι σημαντικό να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο πρώτα απ' όλα δίκτυα που θα συνενώνουν όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και σε διεθνές επίπεδο έτσι ώστε να επιτευχθεί ο απότερος στόχος δηλαδή αυτός της καλύτερης αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεως και εν τέλει της επίτευξης αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, δούμε τι κάνει ο καθένας σε εθνικό επίπεδο, να δούμε πώς μπορεί να συνδυαστεί σε διεθνές επίπεδο ε, αυτή η προσπάθεια. Εμείς έχουμε ένα γενικό ε, διευθυντή ε, ο οποίος ε, ήρθε στο Υπουργείο Εξωτερικών ε, πριν από τρία χρόνια. Έχει έναν πολύ μακρόσυρτο τίτλο, αλλά υπάρχει και λόγος πίσω από αυτό το μακρόσυρτο τίτλο αυτής της θέσης, γιατί, γιατί πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών στη Γερμανία τουλάχιστον ε, είναι αρμόδιο και για την αποτροπή κρίσεων και για τη σταθεροποίηση και για την οικοδόμηση ειρήνης και για την ε, διαχείριση των συγκρούσεων. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία στη θέση του Γενικού Διευθυντή και βεβαίως και ο απαραίτητος προϋπολογισμός και επιχειρησιακά λοιπόν αυτή η διεύθυνση είναι αρμόδια ε, και ε, αυτή η συγκεκριμένη ε, μονάδα μέσω του, της κεντρικής της, του κεντρικού τμήματος αλλά και κάποιων περιφερειακών γραφείων προσπαθεί να επιλύσει συνολικά τα ζητήματα. Πριν από τρία χρόνια καθίσαμε ε, γύρω από ένα τραπέζι και είδαμε τις ε, δυνατότητες διαμεσολάβησης, το ρόλο που μπορεί να παίξει η Γερμανία ε, σε τέτοιες περιπτώσεις, πώς, το ρόλο που θα θέλαμε να παίξει η Γερμανία σε τέτοιες περιπτώσεις. Τρία χρόνια μετά λοιπόν, τώρα, έχουμε Έχουμε δημιουργήσει ε, καλά ε, λειτουργούσες διεθνείς διασυνδέσεις, ε, σωστές διασυνδέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε 40 projects τα οποία υποστηρίζει η Γερμανία στον τομέα της διαμεσολάβησης ε, και ε, βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ε, αυτό δεν το κάνουμε έτσι ώστε να επιβραβευθούμε με το βραβείο Νόμπελ ή κάποιο άλλο για την ειρήνη αλλά θέλουμε, το κάνουμε για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ειρήνευσης, τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την ειρήνευση. Ε, δουλεύουμε με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά όχι μόνο και αποκλειστικά. Προχωράμε και σε διμερείς ε, διαδικασίες. Ε, δίνουμε και οικονομική υποστήριξη, τεχνογνωσία, οποτεδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε και βεβαίως οποτεδήποτε και οπουδήποτε η Γερμανία εμπλέκεται ε, σε διαδικασίες διαμεσολάβησης θα συνεχίσουμε τις διαδικασίες αυτές, τις προσπάθειες αυτές. Ε, δημιουργούμε ε, εταιρικές σχέσεις διότι πιστεύουμε ότι η διαμεσολάβηση είναι ένα εργαλείο αλλά είναι ένα σημαντικό εργαλείο όχι μονάχα για τη διαχείριση ή την επίλυση κρίσεων, αλλά και όσον αφορά την πρόληψη κρίσεων. Η αποτροπή, η διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο αποτροπής σε κρίσεις ή σύγκρουσης. Και γνωρίζω ότι εσείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εκπρόσωποι πολιτικών ε, κομμάτων, ε, μπορείτε να παίξετε σημαντικό ρόλο στην διαμεσολάβηση και εργαλειο αποτροπης σε κριση η συγκρουση και γνωριζω οτι εσεις ως μελη του ευρωπαικου κοινοβουλιου ως εκπροσωποι πολιτικων κομματων μπορειτε να παιξετε σημαντικο ρολο στην διαμεσολαβηση και το κάνετε, γιατί ε, πολλές είναι οι πρωτοβουλίες οι οποίες ξεκινούν είτε από το Κοινοβούλιο είτε από τα κόμματα. Συνεργασίες δε, μεταξύ πολιτικών κομμάτων μπορεί να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτά ήθελα να σας πω και ολοκληρώνω λοιπόν την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κιούνιχ, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Στέφανο Τόματ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνετε να παραστώ στην Επιτροπή σας. Να προλάβω και να πω κάποια πράγματα που νομίζω ότι θα είναι δική σας ερωτήσεις επίσης. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Συνολική Στρατηγική που είναι το πλαίσιο για να συζητήσουμε για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στις συγκρούσεις και στις κρίσεις. Αυτή είναι η απάντησή μας στον νέο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις και στις νέες συγκρούσεις που αναδύονται. Γιατί αλλάζει το κόνσεπτ και οι έννοιες που διαδίδονται. Μιλούμε για ανοχή, για ανεκτικότητα, για αντοχή, για σταθεροποίηση. Έχουμε ε, κόμβους ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς. Έχουμε νέες ιδέες που προκύπτουν τα, οι συγκρούσεις είναι πολύ πιο περίπλοκες με πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις από ό,τι πριν. Και όπως είπε και ο κύριος Ρούντικερ, είναι μια, ένας προβληματισμός που έχουμε εμείς στο EU Global Strategy, αλλά το ίδιο κάνουν και άλλοι φορείς και τα Ηνωμένα Έθνη αυτή τη στιγμή προβληματίζονται για το πώς ε, θα γίνει η πρόληψη των συγκρούσεων βασική προτεραιότητα. Η Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη συνεργάζονται ε, για αυτό το έγγραφο «Μονοπάτια για την ειρήνη» Pathways for Peace και αν διαβάσετε το έγγραφο το συμπέρασμα έχει ως εξής οι συγκρούσεις έχουν αλλάξει ως τη φύση τους πρέπει να είμαστε δραστήριοι καθ' όλα τα στάδια των συγκρούσεων και χρειαζόμαστε ολοκληρωμένη ενιαία προσέγγιση είναι το ίδιο ε, με αυτό που λέμε και εμείς και στα κρατη ο προβληματισμός είναι πολύ παρόμοιος για παράδειγμα, οι προνομιακέ σχέσει που έχουμε με τη Γερμανία απορρέουν από το γεγονό ότι η Γερμανία έχει περάσει μια φάση προβληματισμού πολύ σημαντική για τη σημασία αυτή τη ε, έννοια και μέρο του προβληματισμού οδήγησε στη δημιουργία αυτή τη αρμόδια γενική διεύθυνση. και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ξεκινήσει και έναν προβληματισμό με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και αυτό είναι απαραίτητο μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης Βλέπετε ότι έχουμε μπλέξει την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών περισσότερο στον προβληματισμό μας. Έχουμε οργανώσει μία σειρά εκδηλώσεων με την έμπλο. Το European Peace Building Liaison Officer εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η ΕΜΠΛΟ, δηλαδή ο αξιωματικός σύνδεσμος για την οικοδόμηση της ε, ειρήνης και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Το πρίσμα, η δομή δηλαδή που εκπροσωπώ εδώ, είναι απάντηση σε όλα αυτά. Πρίσμα σημαίνει πρόληψη συγκρούσεων, κράτος δικαίου, ολοκληρωμένη προσέγγιση, σταθεροποίηση και διαμεσολάβηση. Θέλουμε να είμαστε ένα κέντρο υποδοχής όλων των διαφορετικών παίκτων και μπλεκόμενων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα κράτη-μέλη, με το Συμβούλιο. Είμαστε όλο και περισσότερο σε επαφή και σε επικοινωνία με το Κοινοβούλιο. Ο Γκέραρντ ο Γκέρχαρντ που βλέπουμε εδώ είναι ο φυσικός ομόλογος μας και συνομιλητής μας. Ξεκινούμε ανταλλαγές ε, ε, βραχίας περίοδου με ορισμένους αξιωματούχους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη δομή και να βεβαιωθούμε ότι, ότι δουλεύουμε μαζί. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε την εντολή των θεσμικών οργάνων, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι επιχειρησιακά είμαστε στην ίδια πλευρά και συντονιζόμαστε επί, του, επί τόπου. Τρεις είναι οι βασικές ομάδες, θέλω να τις αναφέρω όπως και ο Ρούντικερ. Πρώτον, πρόληψη συγκρούσεων. Έχουμε εκπονήσει ένα έγγραφο ιδεών ενοιολογικό που, το συζη... που συζητείται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και εκεί έχουμε διατυπώσει κάποιες ιδέες. Πρώτη ιδέα, να έχουμε πολιτικές συζητήσεις για την πρόληψη των συγκρούσεων. Το βασικό στοιχείο είναι η πολιτική δράση η πρώτερη. Χρειάζεται να υπάρχει πολιτικό βάρος και να ασκηθεί αυτό το βάρος και θέλουμε αυτό να είναι όλο και πιο παρόν ως κατάσταση και ιδέα στο Συμβούλιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων αρμοδίων για τα θέματα πρόληψης συγκρούσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει οργανώσει ένα τέτοιο δίκτυο και η Γερμανία επίσης. Είναι σημαντικό αυτό το δίκτυο για να υπάρχουν συνδέσεις και αρμόδιοι συνομιλητές μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και κρατών μελών. Θέλουμε να έχουμε εσωτερική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλύει τις συγκρούσεις. Για να παρέμβουμε σε μια σύγκρουση πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, πρέπει να ξέρουμε πού πάμε και τι κάνουμε. Και το πρίσμα το ε, χτίζει αυτή την ικανότητα εκ του μηδενός, να την έχουμε εσωτερικά, να μην την αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους, να μπορούμε να κάνουμε ανάλυση των συγκρούσεων εσωτερικά ενδοϊπηρεσιακά. Εμείς ως πρίσμα. Πρίσμα που σημαίνει πρόληψη συγκρούσεων κράτος δικαίου, ολοκληρωμένη προσέγγιση, σταθεροποίηση και διαμεσολάβηση. Τα προγράμματα είναι σημαντικά, οι πολιτικές είναι σημαντικές, πρέπει να τα συνδέουμε. Τα σημεία σύνδεση ε, μεταξύ ε, και διάρθρωση αυτών είναι, ε, πρέπει να τα προστατεύσουμε και να τα ενισχύσουμε. Ένα σημαντικό στοιχείο στην πρόληψη σύγκρουση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι βεβαίω οι εκλογέ. Όπου εσείς ως Κοινοβούλιο έχετε πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε και πώς να το πω, είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στα οποία πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας όταν ασχολούμαστε με την πρόληψη των συγκρούσεων. Ανέκαθεν είναι ακαθόδε ζήτημα οι εκλογές για κάθε κράτος. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, να δουλέψουμε εκ των προτέρων και να συνεργαστούμε και με εσάς. Για πρώτη φορά έχουμε παράσχει, έχουμε δώσει κατάρτιση, εκπαίδευση σε αυτούς που θα είναι μέλη της, ε, ως παρατηρητές της εκλογικής διαδικασίας της Ζιμπάμπουε και συνεχίζουμε και με τα άλλα όταν θα έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Αυτό προκύπτει από την ιδέα που ε, συζητήσαμε με, το, με την κυρία Σάκε, Ευρωβουλευτή, που είχε ασχοληθεί με το θέμα της Κένιας και είχε ανταλλάξει απόψει μαζί μα Για την διαμεσολάβηση να σας πω ότι αναπτύσσουμε αυτές τις ικανότητες στήριξη τη διαμεσολάβησης εντό του πρίσμα και έχουμε τη στήριξη κρατών μελών, δίδουμε εμπειρογνωμοσύνη, τεχνογνωσία στα κρατημέλη και έχουμε και ευέλικτα εργαλεία για να στηρίξουμε τη διαμεσολάβηση και αλλού σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μία σύμβαση πλαίσιο και θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Κοινοβούλιο, γιατί ήταν δική σας απόφαση να μας δώσετε αυτό το εργαλείο της σύμβασης πλαισίου. Είναι μικρός ο προπολογισμό, αλλά μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε άμεσα ε, δραστηριότητε διαμεσολάβηση ή οικοδόμησης της ειρήνη. Σα ευχαριστώ θερμά γιατί το χρειαζόμαστε ιδιαιτέρω. Και ένα άλλο εργαλείο που φτιάχνουμε, που κατασκευάζουμε μαζί με βάση την εφαρμογή του FBI λέγεται Ερμής και μας επιτρέπει να χρηματοδοτούμε διαδικασίες διαμεσολάβησης με τρίτες χώρες και τρίτα μέρη. Ένα παράδειγμα την δημοκρατία της κεντρο, Κεντρικής Αφρικής, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Μια διαδικασία διαμεσολάβησης ξεκίνησε από την Αφρικανική Ένωση που χρειαζόταν βοήθεια, άρα μέσα από συμφωνία πλαίσιο δώσαμε πυρογνώμονα στον πρόεδρο και βοήθησε τον πρόεδρο να μετρά πώς γίνεται η διαμεσολάβηση και με το πρόγραμμα Ερμής χρηματοδοτούμε και στηρίζουμε τις συζητήσεις που εξελίσσονται και είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή. Θα είμαι πολύ σύντομος. Τέλος, το θέμα της σταθεροποίησης αναφέρθηκε. Εδώ έχει προκύψει μια νέα ιδέα, μια νέα έννοια, ένα νέο κόνσεπτ. Σταθεροποίηση είναι το εργαλείο που μας επιτρέπει να προλάβουμε τη σύγκρουση και το ξέσπασμα βίας πριν προκύψει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να αποστείλουμε πυρογνώμονε ειδικού από τα κρατημέλη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτόπου, εκεί όπου μπορεί να προκύψει προκύψει ξέσπασμα βίας για να λυθεί ε, το πρόβλημα πριν. Έχουμε ένα παράδειγμα στο κέντρο του Μαλή. Κάναμε την άσκηση αυτή, το εγχείρημα αυτό και είχε πολύ θετικά αποτελέσματα. Δώσαμε στήριξη στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για να προλάβουν καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε 10 περίπου λεπτά στην διάθεσή μας. Τρεις είναι οι ομιλητές, τέσσερις από ό,τι βλέπω. Καλώς να ξεκινήσουμε. Τρία λεπτά ο καθένας. Η κυρία Πόστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ε, Ευχαριστώ πολύ και για όλες τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ θα είμαι η συγγήτρια για την έκθεση ε, που έχει σχέση με την ε, δημιουργία μηχανισμού εκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση, τη διαχείριση των κρίσεων. Θα είμαι λοιπόν σε επαφή μαζί σας κατά τη διάρκεια αυτές αυτής της Αυτή την εβδομάδα είχα μία συνάντηση με το αρμόδιο γραφείο για την ε, πρόθεση της ειρήνης. Ε, θα συνεχίσω βεβαίω να έχω επαφές μαζί τους ε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Βλέπω ότι εδώ κοντά μας είναι και μία σκιώδη συγγήτρια από τους πράσινους. Μιλήσαμε για διάφορα θέματα έτσι ώστε να υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης ε, για το μέλλον. Μιλάμε για καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, και επίσης και μιλήσαμε και για το εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης, ε, για τη συμπερίληψη περισσότερων γυναικών και νέων και επίσης αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος ε, πολιτικός ε, στόχος. Επίσης, ε, μιλήσαμε για τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις πρωτεύουσε και για όσους εργάζονται επί τόπου. Για την ανάγκη πολιτικής βούλησης να στηριχθεί η πολιτική διαμεσολάβηση, να γίνουν επενδύσεις σε αυτό το θέμα. Μιλήσαμε επίσης και για τις, ε, ε, την διάμεση διαμεσολάβηση μιλήσαμε για την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις ε, διάφορες μονάδες συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης κρίσεων. Ευρύτερα θα το έλεγα αυτό. Συζητάμε, συζητήσαμε για το εμπόριο, για το περιβάλλον και επίσης μιλήσαμε και για την ανάλυση καλών αποτελεσμάτων για να ξέρουμε ε, πώς μπορεί να υπάρξει μια εύρυθμη λειτουργία. Και μιλήσαμε πολύ και για την συμφιλίωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, το να υπάρξει εμπιστοσύνη. Θα είμαι σύντομη. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Και νομίζω ότι κατά τις αρχές Σεπτεμβρίου θα αρχίσουμε να συντάσσουμε την έκθεσή μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να κρατήσω επαφή και με τους δυο σας στο μέλλον. Ξέχασα ένα πράγμα. Μιλήσαμε και για το πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί η δημοκρατία και η αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγάλη χαρά άκουσα για τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρατε και θα συνεχίσω να ρωτάω και κάτι. Μήπως θα πρέπει κάτι τέτοιο να υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είναι μια ερώτηση που απευθύνω και στους δυο σας και να μας ενημερώσετε και για την, ε, τον εκτελεστικό βραχίωνά σας, το ΣΥΦ. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να δουλέψουμε από αυτού εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως οι Γερμανοί μπορούν να εισάγουν αυτή την ιδέα και στο Συμβούλιο. Γνωρίζω ότι ε, αναφέρθηκε παλαιότερα ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει το PESCO Plus ε, στον τομέα της ασφάλειας ε, των ε, πολιτών και ο κύριος Μας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα ειδικό σώμα για την ασφάλεια, τη σταθερότητα. Ήδη το 1994 το είχε πει ο κύριος Αλεξάνδρ Λάγκε και νομίζω αυτά αναφέρονται σε μία μελέτη ε, την οποία την περάσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν την έχετε, αλλιώς μπορούμε να σας τη δώσουμε. Αυτό, ξέρετε, εγώ έρχομαι από τη Σουηδία και επανειλημμένα έχουμε υπογραμμίσει αυτή την αναγκαιότητα στη Σουηδία. Ίσως λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε οι Γερμανοί και οι Σουηδοί σε αυτό το θέμα για να το προχωρήσουμε σε ενωσιακό επίπεδο. Επίσης, έχουμε να μάθουμε αρκετά για την εξωτερική μας πολιτική. Και όταν πρόκειται για την πρόληψη κρίσεων, ε, όταν υπάρχει επιτυχία, πολλοί δεν το συνειδητοποιούν. Γιατί υπάρχουν πολλές επιτυχημένες ιστορίες, αλλά δεν προβάλλονται. Εδώ στο Κοινοβούλιο μιλάμε περισσότερο για πόλεμο, για άμυνα ε, και για την ειρήνη γενικά, αλλά νομίζω ότι ο ευρύτερο στόχος όλων μας είναι η ειρήνη, οποτεδήποτε μιλάμε για την άμυνα και την ασφάλεια. Κάποτε έκανα μία άσκηση, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, να διαβάσει κανείς ένα έγγραφο και κάθε φορά που προσέκρουε τη λέξη άμυνα να την αντικαθιστεί με τη λέξη ειρήνη. Στο τέλος του κειμένου οι λύσεις που προκύπτουν είναι λύσεις διαφορετικές εάν έχει κανείς καρτανού περισσότερο την ειρήνη από την άμυνα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μας αυτή την άσκηση. Δεν έχουμε τρία λεπτά, δυόμιση όχι τρία. Μία σύντομη ερώτηση σχετικά με το εργαλείο σταθερότητας και ειρήνης, γιατί βλέπω ότι σε αυτό το θέμα υπάρχει μία υπαναχώρηση. Θα μπορούσα να σχολιάσω πάρα πολλά, δεν θα το κάνω. Γιατί εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην άμυνα και την ειρήνη. Όσοι έχουν κατά νου την άμυνα έχουν και την ειρήνη. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό που είπε στο τέλος η κυρία Βαλέιρο. Και συγκεκριμένα το γεγονός ε, ότι υπάρχει μία μετατόπιση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση της ασφάλειας. Αυτό σημαίνει και το βλέπουμε ότι υπάρχει απομάκρυνση και από τους αστικούς εισαγωγικά στόχους. Η κυρία Μογκερίνη έχει φέρει στη συζήτηση ένα νέο εργαλείο, ε, το μηχανισμό για την ευρωπαϊκή ειρήνη, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, με συγχωρείτε, European Peace Facility. Αυτό που συζητάμε περισσότερο όμως ε, είναι πώς θα εξοπλιστούν οι χώρες, ε, είναι στρατιωτικός ο εξοπλισμός, ε, το πώς η λέξη εργαλείο θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το μηχανισμό. Και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται λόγος ε, για τον συνδυασμό διαφορετικών εξωτερικοπολιτικών μηχανισμών ή εργαλείων. Ε, θα ήθελα να ε, σας παραπέμψω σε μία γνωμοδότηση του κ. Μπρόκ για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλή αυτή η ανάλυση και λόγω του χρόνου που έχουμε δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Όμως καθίσταται απόλυτα σαφές ότι με το συνδυασμό διαφόρων εργαλείων, γιατί πρόκειται για 20 περίπου μεμονωμένα εργαλεία, ε, πρόκειται για αστικά εργαλεία, εργαλεία πρόληψης, τα οποία πλέον θα καταπέσουν. Ε, γίνεται λόγος για τον έλεγχο των ε, διαφόρων μηχανισμών, ε, τον, την υποστήριξη διαφόρων επιτροπών που θα απαρτίζονται από εμβληματικές προσωπικότητες. Γίνεται λόγος για πάρα πολλά θέματα. Επ' αυτών όλων λοιπόν θα με ενδιέφερε η δική σας η άποψη για το πώς θα γίνουν εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι, ξέρετε, ε, το βαρέλι έχει πάτο. Δηλαδή αυτά που αφαιρούμε από ένα τομέα προφανώς ε, θα λείπουν από έναν άλλον και όλα αυτά σιγά σιγά περιορίζονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, μου είπαν ότι οι διερμηνείς θα φύγουν, η ώρα είναι 12.30. Όσο είναι οι διερμηνείς ε, παρόντες, μπορείτε να μιλάτε τη μητρική σας γλώσσα, αλλιώς θα πρέπει να μιλάτε αγγλικά.